Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε, ότι δεν είμαστε πολλοί. Καλημέρα σε όλους. Δεν έχω ανακοινώσεις για σήμερα το πρωί. Σας καλωσορίζω όλους. Πώς έχει το σημερινό μας πρόγραμμα. Θα σας ενημερώσω σύντομα για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη. Προτού προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, στις 9.30 θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες για πολλά ζητήματα, για πολλές εκθέσεις μέχρι τις 11.00. και συνέχεια θα έχουμε την Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ μαζί μας από τις 11.00 ως το 10.30 και θα μιλήσουμε για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας ανακοίνωσε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είχαμε το χρόνο να τα συζητήσουμε εκτενώς τότε. Ήταν παρόντες πολλοί συνάδελφοι και θα συνεδριάσουμε και σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 5 και από τις 5 και μετά θα έχουμε τις συνεδρίες των συντονιστών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα σκάφη να ψυχής και τα τομικά σκάφη. Χαίρομαι πολύ που είναι μαζί μας ο κύριος Σβάμπα, ένας από τους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Γκέπχαρτ επίσης θα πάρει το λόγο, η κυρία Ρούλη είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Ρέμπο και η κυρία Πέτη Κάινεν επίσης είναι μαζί μας. Την καλωσορίζω. Αν είστε όλοι έτοιμοι. Θα συνημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα σχετικά με το φάκελο αυτό. Η τελευταία εντελεγή απόψεων έγινε πριν από κάποιο καιρό και ουσιαστικά εργαζόμασταν για ένα συγκεκριμένο ζήτημα της πρότασης αυτής προσπαθήσαμε να δούμε αν τα κριτήρια σχεδιασμού για τα σκάφη, για την ε, κατηγοροποίηση των διαφορετικών ε, ειδών σκαφών αναψυχής, αν τα κριτήρια αυτά θα πρέπει λοιπόν να επικαιροποιηθούν, αν θα πρέπει να αποσαφινιστούν και να γίνουν πιο ασφαλή. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να διεξαχθεί μία μελέτη, την οποία την έχετε λογικά όλοι, μια μελέτη όσον αφορά τα σκάφη αναψυχή και τομικά σκάφη. Δεν έχει προβλεφθεί μια επίσημη παρουσίαση από τους συντάκτε της μελέτης. Θα το κάνω εγώ αυτό. Ελπίζω να είχατε το χρόνο να διαβάσετε πάντως τη μελέτη. Πρωτού σας την παρουσιάσω θα σας πω πώ έχουν τα πράγματα όσον αφορά την πρόταση αυτή καθ' αυτή. Μετά την σημερινή ψηφοφορία θα ξεκινήσει η συζήτηση με την Κυπριακή Προεδρία οι οποίοι μου δήλωσαν ότι θα δώσουν προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, θεωρούν ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδο στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Θα συζητήσω λοιπόν μαζί του μετά τη σημερινή μα ψηφοφορία, να δούμε σε ποιο βαθμό ευθυγραμμίζονται οι απόψει μα και στη συνέχεια θα σα ενημερώσω και θα σα πω αν μπορούμε να συμφωνήσουμε τελικά σε πρώτη ανάγνωση. Αυτή θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Το ζήτημα είναι ακόμα ανοιχτό και θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τη φάση αυτή των επαφών προτού φτάσουμε στις θερινές διακοπές. Θα ήθελα να έχουμε μία βάση για να ξεκινήσουμε τις πραγματεύσεις. Συζητήσαμε τις τροπολογίες την προηγούμενη φορά. Θα ήθελα να σας πω ουσιαστικά ότι είχαμε μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Συμφωνήσαμε για μια σειρά προφορικών τροπολογιών όπου αποκρισταλώνται κάποιε από τι ανησυχίε των σχεδόν εισηγητών. Και ουσιαστικά το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η κατηγορία σχεδιασμού, το μόνο εκρεμέ ζήτημα. Ένα εμπειρογνώμονα από τη Γαλλία, ο κύριο Κοχρίλ, είναι αυτό ο οποίο έγραψε τη μελέτη. Είναι διευθυντή του ICNN, η Γαλλική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των σκαφών και ο ίδιος έχει εργαστεί στην κατασκευή σκαφών. Θεωρώ λοιπόν ότι η μελέτη είναι πολύ καλή, πολύ σαφής και ουσιαστικά βασίστηκε σε μία περίληψη που εμείς του δώσαμε. Θέλαμε ουσιαστικά να δούμε αν οι δικέ μα προτινόμενε τροπολογίε όσον αφορά την αλλαγή των κατηγοριών σχεδιασμού, που ουσιαστικά απομακρύνονται από τι αρχικέ τροπολογίε, ε, συγγνώμη, από τι αρχικέ κατηγορίε σχεδιασμού και ουσιαστικά από την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στι κατηγορίε σχεδιασμού και την προτινόμενη χρήση των σκαφών. Θέλαμε αντικειμενικά κριτήρια που θα έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δύναμη του ανέμου και το ύψο των κυμάτων. ότι περιλαμβάνονται τα κριτήρια αυτή τη στιγμή, στα κριτήρια τα οποία εφίστανται, θεωρούμε ότι δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις σχεδιασμού των σκαφών και πολλές φορές οδηγούν σε λανθασμένη κατηγοριοποίηση και πολλές φορές και οι ίδιοι δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να επιλέξουν ένα σκάφος. Ο, κύριο, ο κύριος Κόχελ, στην μελέτη που έκανε και στην ανάλυση που έκανε της κατάστασης, κάνει τις εξής ε, βασικές συστάσεις. Μας λέει ότι αν ε, απομακρύνουμε τον, ε, το σχετισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον σχεδιασμό του σκάφους και την προτινόμενη χρήση, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε πιο αντικειμενικά, πιο κατάλληλα κριτήρια, όπου θα ευθυγραμμίσουν περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα τα οποία ισχύουν. Νομίζω λοιπόν ότι τα κριτήρια αυτά είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την ποιότητα της κατηγοριοποίησης και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προτείνουμε τα κριτήρια αυτά. Δεν προκαταβάλω αυτή τη στιγμή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια σχετική πίεση. Για ποιο λόγο τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όπως μας λέει ο συντάκτης της μελέτης, και γνωρίζετε επίσης και την εμπειρία που έχει, αντίξωες συνθήκες μπορούν να προκύψουν οπουδήποτε τελικά. Ακόμα και πολύ κοντά στις ακτές μπορεί να προκύψουν πολύ ισχυροί άνεμοι και σε ορισμένε περιπτώσει, ακόμα και στα μέσα του ωκεανού, μπορεί να έχει κανεί πιο ευνοϊκέ συνθήκε ανέμου. Επομένω, οι κατηγορίε σχεδιασμού δίνουν την εντύπωση ότι όσο πιο μακριά κανείς βρίσκεται από την ακτή, τόσο πιο αντίξωε είναι οι καιρικέ συνθήκες. Επίσης μας λέει ότι οι κατηγορίες σχεδιασμούς δεν βοηθάνε τους καταναλωτές να καταλάβουν τις πραγματικές ε, ικανότητες, δυνατότητες κάθε σκάφους. Οι φυστάμενες κατηγορίες δεν επιτρέπουν στον καταναλωτή να κάνει την διάκριση αυτή. Επομένως κάποια σκάφη τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν κύματα και ανέμους της κατηγορίας Β στο ανοιχτό πέλαγος, ενδεχομένως να μην έχουν τα απαραίτητα κριτήρια για να κάνουν κάποιο πολύ μεγάλο ταξίδι, ακριβώς επειδή δεν έχουν την απαραίτητη χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων κτλ. Επίσης, κάποιοι θαλαμιγοί ή μηχανοκίνητα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίσως στα στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς όμως να τα αποκρίνονται πραγματικά στα κριτήρια για, τον, για την ισχύ του ανέμου ή για το ύψος των κυμάτων. Ο συντάκτης επίση της μελέτης κάνει κάποιες άλλες συστάσεις που πιστεύω ότι είναι σημαντικές. Αν δείτε τον πίνακα τον οποίο έχει ενσωματώσει στη μελέτη του, αν δείτε τον αριθμό των σκαφών που έχουν εγκριθεί για κάθε κατηγορία, βλέπετε τελικά, και ενδεχομένως αυτό να σας κάνει εντύπωση, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη τα οποία έχουν κατηγοροποιηθεί στην κατηγορία εκείνη για την παράκτια ναυσιπλοεία. Ουσιαστικά μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες υποκατηγορίες σε αυτή την κατηγορία προκειμένου να κάνουμε μια καλύτερη διάκριση των σκαφών και προκειμένου να δοθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας στις ε, κατηγορίες αυτές όπου ξέρετε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός σκαφών που ε, χρησιμοποιούνται και αγοράζονται. Έχει γίνει και μία πρόταση για μία ρήτρα αναθεώρηση στα πλαίσια των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει για την αλλαγή των κριτηρίων σχεδιασμού. Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αυτά ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση σε δύο χρόνια, προκειμένου να δούμε αν θα πρέπει να προσθεθούν επιμέρους κατηγορίες. Και αυτές οι επιμέρους κατηγορίες θα μπορούσαν να ενσωματώσουν, καθώς επίσης και να ενσωματώσουν τις απαιτήσει για, τα... για τις εκπομπές καυσίμων, τις οποίες έχουμε προτείνει. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το περιλάβουμε αυτό στα πλαίσια μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Γιατί ούτως ή άλλως προβλέπεται να, να αναθεωρηθεί η οδική αυτή, προκειμένου να ενσωματωθούν πιο αυστηρά κριτήρια εκπομπών για τους μικρότερους κυρίως κινητήρες και ενδεχομένως τη χρονική εκείνη στιγμή που θα γίνει αναθεώρηση θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κοινέ υποκατηγορίε για τα νέα σκάφη, τι νέε κατηγορίε δηλαδή που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Βάσει λοιπόν τη ε, μελέτη αυτή που έχουν βγει και οι σα προτείνω να εγκρίνουμε σήμερα τι τροπολογίε που έχω υποβάλει, που θα δημιουργήσουν τι νέε κατηγορίε σχεδιασμού και εφόσον εγκρίνουμε αυτέ τι κατηγορίε σήμερα, θα μπορέσουμε βάσει αυτή τη τροποποίηση να ξεκινήσουμε και συζητήσει με το Συμβούλιο. Για τα υπόλοιπα σημεία συζητήσαμε τους οικειώδεις ηγητές, συζητήσαμε τις υπόλοιπες τροπολογίες που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Μετά την παρουσίαση αυτή μπορώ να δώσω λοιπόν το λόγο στους οικειώδεις ηγητές για να έχω και τη δική τους άποψη για την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σβάμπ, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλή ε, συνεργασία και την εξαιρετική παρουσίαση που κάνατε μόλις. Ε, των όσων συζητήσαμε και στο Στρασβούργο με τους Ε, λίγα έχω να προσθέσω γιατί, γιατί μελέτη συμφωνήσαμε, έχουμε συναντήληψη νομίζω και με τις άλλες πολιτικές ομάδες, γι' αυτό για τις κατηγορίες σχεδιασμού και για τα διαδικαστικά δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα. Πιστεύω επίσης ότι και όλες οι τροπολογίες επί της ουσίας είναι σε καλό δρόμο για συμβιβασμούς Οπότε δεν υπάρχουν και τίποτα τρομερά σημαντικά πράγματα για να επεκταθώ σε λεπτομέρειε. Λείπει τώρα ο συνάδελφος μάντερ, γιατί είναι η μόνη τροπολογία ε, που έχει ίσω κάποια σημασία για τα σκάφη. Προτείνει η εναρμόνιση να γίνει και στις άδειες ε, ε, οδήγησης. Θετικό είναι γιατί ασχολούμαι και εγώ τεχνικά Δεν θέλω να σας ξαναδηγηθώ την ιστορία, τη γνωρίζετε. Αλλά δεν μπορεί να αναφέρεται αυτό το θέμα για τα διπλώματα στην νομοθεσία ε, να είναι για τις κυβερνήσεις μια σύσταση για τους ερασιτέχνες ε, εκείνους που έχουν σκάφη αναψυχής. Ελπίζω τελικά να συμφωνήσουμε. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλή η μελέτη και κρίμα που χρειάστηκε ε, τόσος χρόνος, μάλλον κρίμα που δεν έχουμε τόσο χρόνο και τόσες τεχνικές λεπτομέρειες σε όλα μα τα θέματα για να ασχοληθούμε. Εδώ είναι πολύ υψηλή ποιότητα τη μελέτη αυτή. και Καλό θα ήταν όλοι οι συμμεθέτες που αναθέτουμε στο Κοινοβούλιο που κοστίζουν το ίδιο να έχουν και την ίδια ποιοτική απόδοση. Αυτή είναι μια ευχή που σα εκφράζω. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να ξεκαθαρίσω το εξή. Γιατί κι εγώ ερασιτεχνικά έχω σκάφος αναψυχή. Δεν έχουν καμία σχέση εδώ τα διπλώματα. Ε, γιατί υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εγώ χαίρο πολύ ε, που μπορώ να κυκλοφορώ στα γαλλικά κανάλια χωρίς δίπλωμα ε, χειριστού τέτοιου σκάφους, πράγμα που στη Γερμανία δεν θα επιτρεπόταν. Και δεν θέλω τώρα να δώσω εξετάσεις για να πάρω δίπλωμα χειριστού σκάφους για τα κανάλια, τα εσωτερικές πρώτες οδούς. Καλή πρόταση για τις κατηγορίες ε, σχεδιασμού και η μελέτη. Λέει ο κύριος Ρέπο, τι κοίταξε και τη θεωρεί και εκείνος πολύ καλή και θέλω να το τονίσω κι εγώ, γιατί τόσο συχνά έχουμε πει ε, πόσο κακές είναι οι μελέτες, όχι των δικών μας ανθρώπων, αλλά εξωτερικέ που αναθέτουμε. Λοιπόν, καλό είναι να κάνουμε και επενετικά σχόλια καμιά φορά. Επίση η πρόταση ε, δική σας κύριε Χάρμπορ είναι πάρα πολύ θετική και ο κύριος Ρέπο μπορεί να σας ακολουθήσει σε πολλά από όσα προτείνετε. Και ε, γι' αυτό και αποσύρει και την τροπολογία, του, ε, την υπογραφή του μάλλον για το παράρτημα ένα παράγραφος ένα τα διαβάζω και όλα σημείο α, δεν τα ξέρω εγώ τόσο καλά, γιατί έχει καλυφθεί και ε, δεν χρειάζεται να υπογράφει αυτή την τροπολογία. Ο ίδιος θέλει να ακολουθήσει τη δική σας συμβιβαστική πρόταση για αυτό το θέμα του παρατήματος 1. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάντερς μόλις κατέφθασε. Αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρουλή και μετά σε εσάς. Ich kann mich wieder sehr kurz... ε, πολύ σύντομη θα είμαι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω κύριε Χάρμπερ ε, για την καλή συνεργασία και ήταν πολύ διδακτικό για μένα γιατί δεν ξέρω πώς σκάφη. Ε, ποτέ ε, ούτε αδειοδήγηση έχω, ούτε έχω ανέβει σε τέτοιο σκάφος αναψυχή στη ζωή μου. Ε, είμαι στεριανή, <laughs> μη μου λέτε για καράβια. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας δίνει ο κύριος Χάρμπορ και μας διαφωτίζει και χαίρομαι και για τη μελέτη. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτική για τις νέες κατηγορίες και την ταξινόμηση, αλλά με έπεισε η μελέτη η οποία είναι εξαιρετική πραγματικά και πολύ εύκολα μπορεί κανείς να τα διαβάσει, να τα καταλάβει, ακόμα και αν είναι αδαής και άσχετος περί τα θέματα αυτά. Σε μία μόνο ψηφοφορία θα ψηφίσουμε διαφορετικά. Και αυτό αφορά το βιοκαύσιμα. Γνωρίζετε ότι ως πολιτική ομάδα έχουμε ένα ζήτημα εκεί με ε, την παραγωγή καυσίμων από φυτά που καλλιεργούνται, αλλά κατά τα άλλα έχουμε πολύ μεγάλη σύμνοια. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Ήταν φανταστικά ε, όλα. Και επίσης ε, είμαι και ικανοποιημένος με τον τρόπο ε, που αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό που ζήτησα για το δίπλωμα ε, οδήγησης ε, χειριστού. Να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Το συζητήσαμε χθες τους συντονιστές και χαίρομαι που δίνουμε την ευκαιρία τώρα στους Ευρωπαίους να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα σκάφη αναψυχής και να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Θα πάρουμε και τη Χάιντα μαζί μας. Άλλος κανείς? Θα πω στον κύριο Μάντερς ότι χάσατε την είδηση ότι από τους πιο ηγητές σκάφος έχει μόνο η κυρία Γκέπχαρτ. Αλλά δεν θέλει ένα αρμονισμένο δίπλωμα ε, δίγησης όπως προτείνετε εσείς. Λοιπόν, σας το λέω γιατί το χάσατε αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν τα είχα φανταστεί. Δεν μας τα λέτε αυτά κυρία Γκέπχαρτ ότι έχετε και σκάφη ψυχής. Έπρεπε να είχα καλωσορίσει νωρίτερα και ζητώ συγγνώμη που δεν το έκανα το Λουί Φιλίπε Τζεράου που είναι τμήματάρχης αρμόδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Τσάρλ Κόρκ που είναι ε, ε, επίσης αρμόδιος για την πρόταση και συνεργαστήκαμε ε, στενά. Πέντε λεπτά έχουμε μέχρι τις ψηφοφορίες. Θέλετε το λόγο να μας πείτε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος Κατά πρώτον, σε σχέση με τη μελέτη, επιτρέψτε, για, επιτρέψτε μου για να αποφύγουμε κάθε παρανόηση, να πω ότι είμαστε ανοιχτοί στην αναθεώρηση και την ε, ε, επανεξέταση των διάφορων κατηγοριών, εφόσον χρειαστεί προκειμένου να γίνει μια πολύ ε, περιστατωμένη μελέτη αντικτύπου. Έπειτα, το θέμα των κατηγοριών σχεδιασμού συζητήθηκε κατά την προετοιμασία της όλης πρότασης με τους ενδιαφερομένους, με εκπροσώπους των κρατών μελών, εκπροσώπους των αρχών παρακολούθησης της αγοράς, των ε, φορέων τυποποίησης και των φορέων κοινοποίησης. Δυστυχώς, ως προς τη μελέτη, η μελέτη αυτή βασίζεται σε μία παρανόηση. Η παρανόηση αυτή είναι ότι θεωρείται ότι η προτιθέμενη χρήση είναι καθοριστικό κριτήριο για να οριστεί η κατηγορία του σκάφου. Η οδηγία όμω και η πρόταση δεν αναφέρουν την ε, προτιθέμενη χρήση. Έχουμε ένα εργαλείο όμω για να συζητήσουμε την υλοποίηση τη νομοθεσία μα. Η ομάδα τη διοικητική συνεργασία με όλε τι όλες τις ε, αρχέ των εθνικών κρατών μελών όπου μπορούμε να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες του πώς θα υλοποιηθεί ο νόμος. Και βεβαίω τα βασικά κριτήρια για τα σκάφη και τι κατηγορίε του περιέχονται και στον ανάλογο οδηγό. Εκεί θα ενισχυθούν. Uh, so that, is why in the... Γι' αυτό στην έκθεση εκφράζεται μια σχετική έκπληξη ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα μπορεί να ενισχυθούν ή όχι. βεβαίω πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή και τους εκπροσώπου των κρατών μελών αυτά τα κριτήρια, διότι έτσι έχει δομηθεί το σύστημά μας. Και μάλιστα θεωρήσαμε ότι τα πρότυπα που έχουν ήδη καταρτιστεί συμφωνούν με την νομοθεσία. Ίσως πρέπει να αποσαφηρήσουμε και μια άλλη παρανόηση. Δεν είναι το θέμα των εναρμονισμένων ημί προτύπων που θα καθορίσει την ερμηνεία του νόμου. Το αντίστροφο συμβαίνει. Τα πρότυπα και τα εναρμονισμένα ακόμη θα πρέπει να συμμορφούνται με τις απαιτήσει που προβλέπονται από την νομοθεσία. Όπως είπε ευθύ εξ αρχής, δεν έχουμε λοιπόν προβλήματα ώστε να αλλάξουν οι κατηγορίες σχεδιασμού των σκαφών αρκεί να μπορούμε να αποτιμήσουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Είναι αρκετά περίπλοκο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει βέβαια αυτή η αποτίμηση. Και πρέπει να πω ότι επειδή αναγνωρίζουμε τις θέσεις σας ως αυτές όσων συμμετείχαν στη συζήτηση για την προετοιμασία αυτή, αυτής της πρότασης ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαφωνίες μας εκπλήσει λόγω χάρη που στο κείμενο αναφέρεται ιδίως, ότι αφορά η νομοθεσία για τις κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών, αυτό διαφέρει ως διατύπωση από το κείμενο της οδηγίας. Τα έχουμε συζητήσει αυτά όπως είπα με τους εταίρους, τα κάτι μέλη, τα... τους φορείς κοινοποίησης, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Βεβαίως όλες τις συνεισφορές τις θεωρούμε ευπρόσδεκτες. Για τις αλλαγές λοιπόν των κατηγοριών σχεδιασμού θα χρειαστούμε όπως είπα μελέτη αντικτύπου αλλά σαφώς πολύ εμπεριστατωμένη, ενδελεχή εξέταση του θέματος. Και είναι σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε συνένεση, σαφή συνένεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ιδίω του ενδιαφερομένου, του εκπροσώπου των κρατών μελών, και ακριβώς να δούμε τι αλλαγέ είναι δυνατές. ω προ τι τροπολογίες, κατά την προετοιμασία των τροπολογιών εντοπίσαμε κάποια προβλήματα σε σχέση με ορισμένε από τι προτινόμενε αλλαγέ. Τα προβλήματα παραμένουν σε σχέση με τις κατηγορίες σχεδιασμού, σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη και το άρθρο που αναφέρεται στους ναυτιλωμένους έτσι όπως έχει διατυπωθεί απαιτεί διαρκή έλεγχο όλων των ε, μηχανών. Κάποιες φορές όμως είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος του ελέγχου για τις μικρές μηχανές από ότι ίδια η αξία της μηχανής. Έτσι λοιπόν όπως έχει διατυπωθεί το εκτιμώντας αυτό θα παρατείνει την υποχρέωση των κατασκευαστών Ακόμα και για αυτούς που μετατρέπουν τις μηχανές για να προσαρμοστούν ε, στα διάφορα σκάφη. Υπάρχει και μια τροπολογία όπου αναφέρεται ότι οι έλεγχοι για το θόρυβο θα ακολουθούν τα πιστοποιημένα πρότυπα. Όμως αυτά τα πιστοποιημένα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά. Η νομοθεσία βασίζεται στο γεγονός ότι τα πρότυπα δεν είναι δεσμευτικά ακριβώς. Τα εναρμονισμένα πρότυπα προβλέπουν λοιπόν ελέγχους αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να είναι δεσμευτικά. Σας ευχαριστούμε και ευχαρίστως να διευκολύνουμε τους ενδεχόμενους συμβιβασμούς που μπορεί να βρεθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε συνεισφορά μας ζητήσετε. Ευχαριστώ. Okay, well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. λύσαμε αρκετά ζητήματα. Ε, δεν ξέρω θέμα ερμηνεία. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. Ε, όταν θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε θα επανέλθω στην Επιτροπή για να μου δώσουν εντολή να αρχίσω τις διαπραγματεύσεις. Um, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να πει τίποτα άλλο. Προτείνω να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να μαζευτούμε για τις ψηφοφορίες, να ετοιμαστούμε και να ε, ψηφίσουμε πρώτα την οδηγία για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. αντίπατη και Uh, are we ready to vote, everybody? Good morning, everybody. Good. Yes, thank you very much. Thank you. Uh, I have people keep... Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να πω σε όλους όσοι δεν ήταν προηγουμένω εδώ καλημέρα. Συζητήσαμε ένα συνεπαστικό θέμα για τις κατηγορίες σχεδιασμού. Κρίμα που το χάσατε, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να αναπληρώσετε πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και μέχρι να έρθουν ακόμη περισσότεροι, να ευχαριστήσω τον κύριο Ούντερ, ο οποίος ε, θα μας αφήσει δυστυχώς μέλος του προσωπικού. Θα εργαστεί στην ομάδα οικονομικής συνεργασίας στα τέλη Ιουνίου και θα φύγει από κοντά μας. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν για όλη τη σκληρή δουλειά ως τώρα. Είναι πολλά χρόνια μαζί μας εδώ, μεταξύ των μελών του προσωπικού. Σίγουρα όλοι συνεργαστήκατε μαζί του σε κάποια φάση. Και πραγματικά έχεις κάνει πολλή δουλειά για μας και στο Σουηδικό και στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο προσκαλώντας και εκπροσώπους των κοινοβουλίων αυτών εδώ κοντά μας. Λοιπόν, να δούμε καταρχάς την οδηγία για τα σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη. Ε, Επιτροπή Τραν, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 8 καταπίπτει, 40, αποσύρεται μάλλον, 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 και τραν 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ εγκρίνεται 49 και 50 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται 51 αποσύρεται 52 υπέρ κατά εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 και 54 μαζί. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 13 αποσύρεται. 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17 και 18 αποσύρονται. 55 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επιτροπή Μεταφορών 12 υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. NV4, Επιτροπή Περιβάλλοντος 4 επιτροπη Περιπαραντός κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56. Θα την ψηφίσουμε αργότερα την τοπολογία 56 διότι αφορά την ομάδα των κατηγοριών σχεδιασμού. 56 με μια προφορική τροπολογία λοιπόν που θα την παρουσιάσω μετά. 57. Εντάξει όλοι. 57 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58 αποσύρεται. Διότι θα υπάρξει μια νέα τροπολογία που θα αφορά τη ολογική σκέψη και η οποία θα προκύψει αργότερα. Τώρα, για τις κατηγορίες σχεδιασμού που μόλις συζητήσαμε. Θα έλεγα να ψηφίσουμε ομαδικά. 21, 59, 62, 61, 62 και λοιπές. Και αυτό μαζί με τη δική μου προφορική τροπολογία. Για τις νέες κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών λοιπόν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περιλαμβάνονται λοιπόν όλες αυτές τις τροπολογίες και 56, οπότε τώρα προχωράμε στην 60 που καταπίπτει, 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Παραρτήματα. 30 υπέρ κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τρανς, ε, Επιτροπή Μεταφορών 13 υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ξυπνήσει και το μηχάνημα. Υπέρ της Τραν 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35, 34, το αντίστοιχο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 36, αποσύρεται. 66, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 34 καταδιεπτή, 37 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις ατολικές σκέψεις. Τραν 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Επιτροπή μεταφορών 2, τραν 2, 3 συγγνώμη, 3 υπέρ νομίζω υπέρ κατά απορρίπτεται. Τραν 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 3 αποσύρεται και 4 το ίδιο 42 υπέρ κατά εγκρίνεται τραν 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 κατά πίπτη 2 υπέρ κατά εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 26 Προφορική τροπολογία του κ. Μάντερ που την έχετε στην κατάλογο ψηφοφορίων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 28. NV3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 43. Με προφορική τροπολογία. Από τον κύριο Μάντερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43 καταπίπτει, 44 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 αποσύρεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τραν 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίση. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την πρόταση συνολικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται με 30 προς 1. Ευχαριστούμε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους χρήστες καθόλου στην Ευρώπη. Περνάμε τώρα στην κοινωνική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα της κυρίας Χάνσλικ. Πάμε απευθεία στην προφορία. Γι' αυτό δεν είναι εδώ η κυρία Χάνσλικ. Είναι εδώ η κυρία Χάνσλικ. Okay, in the digital agenda. Perfect. Right, let's move on to Mrs. Hanslick's opinion then. Ας περάσουμε στην γνώμη ε, της κυρίας Χάνσλικ. Ένα. Χάνσλικ τη πρωτοβουλία. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Συμβαστική ένα. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 7. Κρύο γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Με διαφορά. Οκτώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8. Νομίζω πρέπει να ξαναρχίσουμε. Κάποιο δυσκολεύεται με τα κουμπιά σήμερα. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία που θα προσθεθεί εδώ την έχετε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. συμμεπεστική 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14. 14. Άρχεται η προφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τρία. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 του κ. Γκρέχ. Υπέρ. Άρχεται η συμφορια μάλλον. The Πέρας. Απορρίπτεται. 15-15. Ισοψηφία. 5, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία για την 30. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε ολοκληρώσαμε με τις τροπολογίες και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Ευχαριστούμε κυρία Χάνσλικ, παρόλο που λείπετε. Πολύ καλά, θα τα παρουσιάσει και στην άλλη αρμόδια επιτροπή. Τώρα έχουμε την έκθεση Weisgerber για την οικοστάθμη των μηχανοκινήτων οχημάτων. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Weisgerber. Ωραία. Περνάμε απευθεία στην πληροφορία, λοιπόν. No, I think by the time we we get on. Right. Okay, let's go. Uh, amendment by the Τρία της εισηγητρίας. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ, εγκρίνεται. 22. Υπέρ,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 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 ως προσθήκη υπέρ, κατά, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, 24. Άρχεται την ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ και 13 κατά. 13 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 26 ε, καταπίπτει. 14. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα προτείνεται να ψηφίσουμε ομαδικά όλες τις αιτιολογικέ σκέψεις. Συμφωνείτε όλοι ωραία. Υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνονται όλα. Πάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία απευθείας. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Για δύο εποχές. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βάιτ Κέρμπερ. Θα περιμένουμε να σας ακούσουμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μπράβο. Και τώρα η έκθεση του κυρίου Ροσφόρ για το πρόγραμμα των καταναλωτών. 2014-2020. Ο εισηγητής. Θέλετε το λόγο. Συζητήσαμε τις κελίες συμβαστικές τροπολογίες χθες με του συναδέλφου οπότε ας πάμε απευθείας στην ψηφοφορία. Can ξεκινήσουμε. Τροπολογία 87 του κυρίου Τρενταφυλλίδη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 κυρίου Ροσφόρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιπρόσθετα έχουμε και προφορική τροπολογία, την οποία τη βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφορίας από τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών. Budget 9, λοιπόν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τζούρι 3 επιπρόσθετη υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 88 πίπτη, γιατί συσχετίζεται με το 87. Περνάμε στην τροπολογία 10 του συγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 11, 15, 47 και 64 από κοινού υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η τροπολογία 89 καταπίπτει. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Περνάμε στη βασική τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Γιούρι 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 93 του συγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η Γιούρι 6. Budget 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 κυριοσφόρ υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 95 του κύριου Γκρέχα υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 95 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Επιτροπή Προπολογισμών υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 96-113 μαζί υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 16 έχει αποσυρθεί και η 48 επίσης. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβασική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 21 και 58 μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 8 γιούρι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 του κ. Λουί Γκρέχ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 23 και 126 μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται και οι δύο. Τροπολογία 107. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Τροπολογία 108. Άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 108. Κάποιος καθυστερεί με την ψηφοφορία, είναι πολύ αργός. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 12 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 24 και 129 μαζί υπέρ, κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 62 επιπρόσθετη υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 128. Οι 25 και 63 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και οι δύο. 109 και 26. Με συγχωρείτε. Η τροπολογία 109 μόνο. Αυτή τη στιγμή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 28 υπέρ. Μάλλον πρέπει να ελέγξουμε για τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 με την προφορική τροπολογία που βλέπετε υπέρ κατά εγκρίνεται η 31 καταπίπτει στην αρχική της μορφή τροπολογία 13 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ κατά εγκρίνεται 32 υπέρ κατά εγκρίνεται 33 άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 33 Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Budget. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36, 38, 43 και 8 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 15 της Επιτροπής Προπολογισμών. Καταπίπτει αυτή η τροπολογία. Το πρώτο τμήμα και περνάμε στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο επιπρόσθετο τμήμα της 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 του κύριου Τρενταφυλλίδη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 111, μάλλον αυτή καταπίπτει. Περνάμε στις 40, 41 και 42. Μάλλον στην 44, υπέρ. Υπέρ για τις 44, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 45, 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50, η 50 έχει αποσυρθεί 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 122 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η αρχική μορφή της 122 καταπίπτει 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127. Άρτη ψηφοφορία για τροπολογία 127. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η αρχική 61 καταπίπτει. Τροπολογία 9 γιουρι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65, 66, 67 και 68 μαζί υπέρ. Μάλλον άρτη ψηφοφορία, συγγνώμη. Άρτη ψηφοφορία για αυτές τις τέσσερις τροπολογίες. Πέρας. Απορρίπτονται. 16 κατά 15 υπέρ. Τροπολογία 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι τροπολογίες 73 και 74 από κοινού με την προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε. Νομίζω ότι ο ε, μπλοκ θα τις ψηφίσουμε υπέρ, κατά. Εγκρίνονται και οι δύο. Οι 73 και 74 καταπίπτουν. Περνάμε τώρα στην τολική σκέψη 75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απο... εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 του κύριου Λουί Γκρέχ με τις προφορικές τροπολογίες υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η αρχική 76 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 επιπρόσθετη άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 78. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, Γιούρι, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 4. Τις επιτήσεις προπολογισμών υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 83 μάλλον καταπίπτει 83, συγγνώμη. Περνάμε στη συμβασική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 85. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 85. Πολύ ωραία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 προς 12. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Budget υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, δεν υπάρχει για αποχές. 7 της Επιτροπής Προπολογισμών. Άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ευθυγραμμίζεται με τις άλλες ψηφοφορίες. Περνάμε στην 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 3. Εδώ πέρα έχουμε κατά τμήματα. Η Άλντε μας το έχει στήσει αυτό. Πρώτο τμήμα. Άρτε ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο σύνολο της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 ψηφί υπέρ, εγκρίνεται μία ψήφος κατά και μηδέν αποχές. Okay. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ροσφόρ. Τώρα εσείς θα κληθείτε να υπερασπιστείτε αυτή την πρόταση. Παρακαλώ μην φεύγετε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι για εντολές διαπραγμάτευσης πρέπει να συμφωνήσουμε το κείμενο για δύο προτάσεις και χρειάζομαι τη πλήρη υποστήριξή σας στην ψηφοφορία παραμείνετε και είναι και από ευγένεια και προς τον εισηγητή. Εισηγητές, ο κύριος Μπίλαν, θέλει να πει τίποτα για το θέμα σας. Ε, σύστημα προφόρησης για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι διαπραγματεύσεις ε, ολοκληρώθηκαν με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρκετά καλό αποτέλεσμα και θετική απάντηση από πλευρά του Συμβουλίου και συνιστώ πραγματικά στην Επιτροπή την υπερψήφιση του κειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους και οδησυγητές γιατί κάνατε πολλή δουλειά. Λοιπόν, καλό θα ήταν να εγκρίνουμε τη θέση αυτή και επίσημα και τυπικά. Δεν ξέρω, χρειάζεται και ηλεκτρονικά. Ποιοι είστε υπέρ ε, της έγκρισης ε, της θέσης της συνδιαλλαγής για να πάει στην Ολομέλεια. Κατά αποχές. Δύο αποχές. Θέλετε ηλεκτρονικά για να υπάρχει αποτέλεσμα και ίχνος να αφήσουμε. Ωραία, ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία. Vote electronically, so we have clear... Έχουμε σαφή καταγραφή έτσι. Συγγνώμη, Κρίστη. Μην βγάζετε τις κάρτες σας. Είναι ε, και για τα πρακτικά. Για να έχουμε μια σαφή ψηφοφορία και ένα αποτέλεσμα. Ah, okay. The vote is closed. Πέρας. 24 υπέρ, κανείς κατά δύο αποχές. Κυρία Τούρεν, αν εσείς ψηφίζετε υπέρ, γιατί δεν έχετε κάρτα. Α, έχετε, εντάξει. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η επόμενη ε, έκθεση είναι της κυρίας Κόμη για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Κυρία Κόμη, θέλετε να πείτε δύο λόγια πριν εγκρίνουμε και τη δική σας θέση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά και τους σκιώδεις εισηγητές. Ήταν μακρά ε, όλη προσπάθεια και περίπλοκη αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε μια τελική συμβαστική πρόταση. Θα ζητούσα λοιπόν να προχωρήσουμε βάσει αυτής και να φτάσουμε με αυτή και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι ψηφίζουμε τυπικά για την πρόταση της κυρίας Κόμη για να εγκρίνουμε το πακέτο για την τυποποίηση, όπως το διαπραγματεύτηκε με το Συμβούλιο. Άλλος κανείς. 25 κάρτες βλέπω. Ανεβαίνει. Σιγά σιγά. Η κυρία Κόνη θα θέλει φαντάζομαι τη μέγιστη υποστήριξη. Άλλος. Φέρας. Ε, σιγά σιγά αυξάνονται. Ορίστε. 100% 27 όλοι υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Good. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τέλειωσε τόσο γρήγορα η ψηφοφορία. Είχαμε προβλέψει πολύ περισσότερο ε, από ώρα. Ο κύριος Μπαρνιέ δεν θα έρθει πριν τις 11. Ε, μικρό ή μεγαλύτερο διάλειμμα για καφέ. Μην φύγετε, να έρθετε στις 11 γιατί έχουμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρνιέ. Ζητώ συγγνώμη. Ήσασταν τόσο αποτελεσματικοί στις ψηφοφορίες, την άλλη φορά θα βρούμε κανένα θέμα να προσθέσουμε. Παρακαλώ να ξανάρθετε και ελπίζω να ξανάρθετε στις 11. 11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 Ας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 Κυρίες και κύριοι, Κατήστε παρακαλώ. Uh, um- λοιπόν, θα ήθελα και πάλι να καλημερίσω το κοινό μας και στο διαδίκτυο. Όπως γνωρίζετε ψηφίσαμε τόσο γρήγορα που τελειώσαμε νωρίτερα και κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Χαίρομαι που βλέπω τόσους πολλούς συναδέλφους εδώ παρόντες. a um, και όπως πάντα με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Επίτροπο κύριο Μισελ Μπαρνιέ Αρμόδιο για την εσωτερική αγορά. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψή του εδώ σήμερα, διότι οι περισσότεροι πιστεύω συμμετείχαμε την περασμένη εβδομάδα στη συζήτηση στο Στρασβούργο που παρουσίασε δύο πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για την οδηγία για τις υπηρεσίες, τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την πράξη ε, της ενιαίας αγοράς. Όπως γνωρίζετε, πέτυχε πάρα πολύ και το ψήφισμά μας στην Ολομέλεια. Ψηφίστηκε από 550 και πλέον βουλευτές. Θέλω να πω σήμερα το πρωί στον Υπουργό, στον Επίτροπο, ότι η Επιτροπή μας ενέκρινε ε, τη συμφωνία με το Συμβούλιο για ε, την τυποποίηση από τους 12 μοχλούς όπως ονομάζονται που πρέπει να συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο είναι ο πρώτος που εγκρίνεται. Οπότε εμείς όχι μόνο προωθούμε την πράξη ενιαίας αγοράς αλλά περάσαμε και το πρώτο μοχλό. Έχουμε και άλλους μοχλούς που ακολουθούν, άλλους 11. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και χαίρομαι που είναι όλοι εδώ παρόντες θα ήθελα να απευθυνθώ στον Ταμιά Μπατ και να το συγχαρώ για την εκλογή του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Λυπούμαστε πάρα πολύ που θα μας φύγει, διότι ήταν πάρα πολύ ενεργό μέλος στην Επιτροπή μας και δραστήριο. Συγχαρητήρια για την εκλογή σου και στο καλό. Ίσως είναι η τελευταία φορά που συμμετέχεις εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα όσα έκανες στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον Μισό Μπαρνιέ και μετά έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση μέχρι τις 12.30. Οπότε θα έχετε όλοι ερωτήσεις, φαντάζομαι θα τις ομαδοποιήσουμε ανά δύο, τρεις και θα έχετε την ευκαιρία να γίνει συζήτηση με τον Επίτροπο. Καλώς όρισατε και πάλι, σας δίνω αμέσως το λόγο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Χάρμπορ για την ε, υποδοχή σας και για τη μόνιμη πρόσκληση που έχω και χαίρομαι ε, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλογο άμεσο όσο και σε βάθος όπως σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, για την απόφαση που επιβεβαιώσατε για την πρώτη ε, πρόταση κλειδί, τον πρώτο μοχλό με την τυποποίηση για την πρώτη ενιαία πράξη. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας λόγος, μια διανοητική εφεύρεση πράξη για την ενιαία αγορά είναι συγκεκριμένες προτάσεις μια σειρά προτάσεων που θα αλλάξουν το ίδιο το οικοσύστημα, για να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών. Ελπίζω στη γραμμή αυτή, μετά την πρώτη επιτυχία που συνεισέφερε πολύ το Κοινοβούλιο, την άλλη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα έχουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν και μια δεύτερη μείζωνα επιτυχία με τη δημιουργία επιτέλους ε, του ε, ενιαίου Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρυσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ρυθμίζοντας το τελευταίο θέμα που εκκρεμεί ως ε, προς την έδρα του δικαστηρίου. Παρίσι, Μόναχο και Λονδίνο ερίζουν. Και εγώ να συγχαρώ τον Ταμιά Αμπάτ που δυστυχώς θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευτυχώς από την άλλη σκοπιά θα ενταχθεί ε, στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου θα δώσει ε, μια επιπλέον ευρωπαϊκή πινελιά σε μια γαλλική συζήτηση που τη γνωρίζω πολύ καλά και είναι πάντα πάρα πολύ εθνοκεντρική, γαλλογαλλική. Καλό είναι λοιπόν και στην Εθνοσυνέλευση και στο Γαλλικό Κοινοβούλιο να έχουμε μια αρμόδια ευρωπαϊκή φωνή, όπως είναι εκείνη του κυρίου Μπάντου. Πρόεδρε, θυμούμε τη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο πριν από λίγες μέρες. Εκεί είχα την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο πιστεύω και μας υποχρεώνει να ε, φροντίζουμε για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η μεγάλη εσωτερική αγορά σε αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε είναι το πρώτο ενδεχόμενο θύμα της κρίσης και της επιστροφής στον προστατευτισμό γιατί αισθανόμαστε ότι ανεβαίνει αυτό μαζί με την κρίση σε πολλές χώρες. Είναι ένα αντανακλαστικό, εθνικό, για να μην πω καμιά φορά και εθνικιστικό, που πάντα στρέφεται κατά της Ευρώπης και υπέρ του προστατευτισμού. Ταυτόχρονα όμως η εσωτερική αγορά είναι η πρώτη ευκαιρία, το πρώτο μας ατού για να βγούμε από την κρίση και να βρούμε το δρόμο της ανάπτυξης. Εξού και η κοινή μας υποχρέωση να αναζητήσουμε αυτά ε, τα δύο, τρία, 4% ποσοστιαίες μονάδες μεγέθυνσης της οικονομίας το περιμένουν και επιχειρήσεις και οι πολίτες. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα ένα-δύο λεπτά να αναφερθώ σε κάτι που μου έκανε εντύπωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά που είπε ο κύριος Χέλμερ, έδωσε κάποια αριθμητικά στοιχεία που είναι λανθασμένα. Εγώ δεν θέλω να κάνω πολεμική αντιπαράθεση εδώ, δεν είναι του χαρακτήρα μου, αλλά ορισμένα στοιχεία για την προστιθέμενη αξία της εσωτερικής αγοράς χρειάζονται. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2008, πριν από λίγα χρόνια, το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών ήταν 2,13% επιπλέον από όσο θα ήταν χωρίς να έχουμε εσωτερική αγορά ή 233 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ανακάτοικο συν 500 ευρώ χάρη στην εσωτερική αγορά. Αντί να ήταν ο καθένας στη γωνιά του με την εθνική του εσωτερική αγορά, ο καθένας για τον εαυτό του. Άλλο στοιχείο αριθμητικό που θα ήθελα να σας αναφέρω. Ε, την τελευταία 20 αιτία από τότε που ιδρύθηκε η εσωτερική αγορά, το ενδοκινοτικό εμπόριο, χάρη στην εσωτερική αγορά, αυξήθηκε από 800 δις ευρώ το 92 σε 2,8 δις το 2011. Καταλαβαίνετε, οι χώρες, 27 ε, σημερινές μεταξύ τους, από 800 δις σε 2,803. και το διασυνοριακό εμπόριο ήταν μόλις 12% το 1992. Επίσης, ε, θέλω να θυμίσω ότι η εσωτερική αγορά σημαίνει ε, συγκεκριμένες πρόοδους. Από το 1998 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί στο 1 τρίτο το κόστος των τηλεφωνικών ε, συνδιαλέξεων. 93% έχει μειωθεί σε σχέση με το 2005 το να δέχεσαι ένα τηλεφώνημα στο εξωτερικό. Δεν είναι ε, σοβαρό ούτε σωστό να λέγεται αυτό που ακούστηκε στην Ολομέλεια της προάλλες, ότι το κόστος της ενιαίας αγοράς ε, υπερβαίνει το όφελος ή την προστιθέμενη της αξία. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας ε, αφοσιωμένοι στο δρόμο αυτό της ευάνθησης της ενιαίας αγοράς και στις χρηματαγορές που ενδιαφέρουν πολύ και τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται μέγας λόγος τώρα για την ανάπτυξη, γιατί ο κόσμος αυτό περιμένει, που ανησυχεί ή που ε, έχει ε, οργιστεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για λιτότητα, για διαχείριση, για δικυβέρνηση. Μπορεί να χρειάζεται εξυγίανση και σταθεροποίηση του προπολογισμού, αλλά πρέπει να ξαναβρούμε και το δρόμο της ανάπτυξης. Την άλλη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πέρα από κάποια συγκεκριμένα σχέδια που ελπίζω να λάβουν ε, σάρκα και ωστά, τα ομόλογα έργων, τουλάχιστον η πρώτη φάση ελπίζω, τα project bonds, η καλύτερη χρήση των διαθωτικών ταμείων, ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εξ όσων γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφανθεί και για μια σειρά μέτρων που θα επιφέρουν ε, ταχεία κέρδη, ωφέλη για την ανάπτυξη, τα λεγόμενα quick wins. Σύντομα, θα ήθελα να αναφερθώ στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να επιμείνω γιατί τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και στη συνέχεια συγκεκριμένα μέτρα και να κάνω και ένα απολογισμό της πρώτης πράξης για την ενιαία αγορά. Πρώτος στόχος, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί πέρα από τα νέα έργα και τα σχέδια και πριν από τα νέα σχέδια θα πρέπει να ελοποιήσουμε ε, ε, σωστά τα ε, όσα ήδη έχουμε αποφασίσει να λειτουργεί σωστά η νομοθεσία και ιδιαίτερα η οδηγία για τις υπηρεσίες και γνωρίζουμε τη σημασία. Θα σας διανύμω μερικά έγγραφα και μεταξύ αυτών έναν πίνακα όλων των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τρόπος με τον οποίο καλύπτονται ζήτησα να γίνει το έγγραφο στα αγγλικά, το είχα μόνο στα γαλλικά, για να ε, βλέπετε αναϋπηρεσία πώς καλύπτεται η κατάσταση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 95% των ε, υπηρεσιών καλύπτονται ήδη ε, από κοινοτική νομοθεσία εκτός από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα επέγνια στο διαδίκτυο θα πρέπει να δούμε πώς μέσα σε 5 με 10 χρόνια μπορούμε να κερδίσουμε 0,8 έως 1% επιπλέον στην ε, μεγέθυνση της οικονομίας. Το κείμενο λοιπόν που σας παρουσίασα προσωπικά στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα θα ε, είναι λειτουργικό, επιχειρησιακό, πάρα πολύ συγκεκριμένα, με αυστηρή πολιτική ε, σε περίπτωση παραβίασης, μηδενική ανοχή όταν παραβιάζεται σαφώς η οδηγία για τις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην καλύτερη λειτουργία των ενιαίων θηρίδων. Επίσης θέλω να ε, βελτιστοποιηθεί η χρήση τόπου διαφόρων μέσων της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό κάναμε δοκιμές ε, απόδοσης ανάμεσα στις διάφορες οδηγίες για τις υπηρεσίες, για τα επαγγελματικά προσόντα ή την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Διάδραση μεταξύ λοιπόν των ευρωπαϊκών κειμένων για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κινητικότητα, στις ασφάλειες ή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, θα ήθελα να είναι εγγυημένα τα ωφέλη των οδηγιών για τους καταναλωτές προλαμβάνοντας τις διακρίσεις που γίνονται αυτό τον καιρό ε, βάσει εθνικότητας ενός καταναλωτού ή ε, τόπου διαμονής του οδηγία λοιπόν για τις υπηρεσίες, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Από την άλλη υπάρχει και η καλύτερη διακυβέρνηση της εσωτερικής ενίας αγοράς και ξέρετε ε, αυτό που με δεν είναι μια τεχνοκρατική θεώρηση. Αλλά εάν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, αυτό είναι επιζήμιο για την ίδια τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και επίσης προκαλεί και ε, στρεβλώσεις, διαταραχές. Έχετε εργαστεί πολύ η κυρία Κανιέτ, ο κύριος Μπούσου, η κυρία Μπάστο σε αυτά τα θέματα και χαίρομαι που σε συνέχεια του ψηφίσματος που εγκρίνατε την περασμένη Πέμπτη θα ε, οριστεί και ένα νέο εισηγητής, ο κύριος Ανδρέας Φαμπ και θα μπορέσει να εργαστεί με πολύ μεγάλη προσοχή ε, για όλα αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε η εσωτερική αγορά και τα κείμενά μας να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα όταν ομιλούμε για εσωτερική αγορά. Πρότεινα στον Όλυ Ρεν, τον συνάδελφό μου, και συμφώνησε, γιατί είναι επιφορτισμένο με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ζήτησε αυτό να μην είναι αμυγό δημοσιονομικό ή οικονομικού συντονισμού εξάμεινο, αλλά και ένα εξάμεινο που θα προλαμβάνει τι εξελίξει στην ανταγωνιστικότητα και στη μεγέθυνση τη οικονομία παντού στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή, να υπάρχει και ένα κεφάλαιο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που να αφορά την ε, ενιαία εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα. Και με benchmarking, δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα εντός της ενιαίας αγοράς ή ακόμα και τις αδυναμίες ε, ως προς την ανταγωνιστικότητα ορισμένων κρατών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκτός από αυτή τη διαχείριση της οδηγίας των υπηρεσιών ή της ενιαίας αγοράς, αποφασίσαμε από κοινού και ήταν σημαντική η δική σας συνεισφορά να δράσουμε συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρώτης ενιαίας πράξης πράξη για την ενιαία αγορά. Τηλεγραφικά να θυμίσω το στόχο μας για διάφορα κείμενα και τον συνολικό στόχο να καταλήξουμε πριν τα τέλη του έτους, αν συμφωνείτε, σε 12 προτάσεις, κλειδιά αυτή η μοχλή, ε, να ε, δοκιμήσουν. Είδαμε την τυποποίηση που πέρασε, ελπίζω τα διπλώματα τεχνία την άλλη εβδομάδα και πριν το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Για τα επαγγελματικά προσόντα και τη σχετική οδηγία υπό την αιγίδα της κυρίας Μπερναντέτ Βερνιό και ημών ε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθεσμίες. Ελπίζω το συντομότερο να εγκριθεί αυτό το κείμενο. Το συζητήσαμε στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ιδέα της επαγγελματικής κάρτας ή ταυτότητας είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται. Βέβαια, απομένουν λεπτομέρειες. Προσωπικά, εγώ δεν είμαι υπέρ ε, της ε, υπόθεσης του πολλαπλασιασμού των opt-out, της αυτοεξαίρεσης γιατί είναι νέος κατακαιρματισμός. Πάντως είμαστε στη διάθεσή σας με τους συνεργάτες μου για να συνεχιστεί η συζήτηση. Δεύτερο θέμα, δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο σεβασμό της εσωτερικής αγοράς και ε, την απλούστευση και την εγκάρσια ε, ε, πολιτική για την έρευνα, το περιβάλλον, την κοινοτομία. Είναι πολύ δραστήριος ο κύριος Μάρκ Ταραμπελά, εισηγητής, και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, οι δημόσιες συμβάσεις είναι κάτι ε, που χρειάζεται απλούστευση οπωσδήποτε, διότι οι διαγωνισμοί θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλη την Ευρώπη. Μία από τις τάσεις μου στη δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά θα είναι ίσως οι ε, ε, ψηφιακοί διαγωνισμοί ε, τις δημόσιες συμβάσεις. Να φύγουμε από τα χαρτιά και να περάσουμε στην ψηφιακή διάσταση. Επειδή είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των προμηθειών στην Ευρώπη. Όχι μόνο θα μειωθεί η γραφειοκρατία έτσι, αλλά οι οικονομίες θα είναι 80 με 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο καταργείται έτσι τόσο διοικητικό κόστος. Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι κάτι που πρότεινε η συνάδελφός μου Νέλη Κρούς. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή των δημοσίων συμβάσεων. Και στη δεύτερη ενιαία πράξη επίσης θα αναφερθώ και ε, στα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τρίτο θέμα. Τρίτο κείμενο και χαιρετίζω το Φιλίπ Ζουβέν που προχωρεί εισηγητής όσο γίνεται να απλουστεύουμε τα κείμενα της Επιτροπής ε, για τις εκχωρήσεις να έχουμε πρόοδο. Ξέρω το χρονοδιάγραμμα αμφισβητείται καμιά φορά, θα πρέπει να υπάρχει μια βάση σαφής για την πλαισίωση ε, των ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα και να εξασφαλίζονται οι επιχειρήσεις που ε, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με εκχωρήσεις, σε παραχωρήσεις ε, κάποιων κλάδων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο της αμοιβαιότητας που πρότεινα με τον συνάδελφο Ντεχούχτ. Είναι ένας μοχλός διαπραγματεύσεων και μας χρειάζεται για να ανοίξουν αγορές κλειστές σε μας. Βλέπε Κίνα αλλά χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη για να αποφύγουμε να εφαρμόζεται το GPA με τρόπο ασυνάρτητο, ασυντόνιστο και διαφορετικό σε διάφορες χώρες μέλη. Ο κύριος Ντοχιούχτ δεν θέλει να κλείσει τις δικές μας αγορές, αλλά να ανοίξουν οι άλλες ε, βάσει αμοιβαιότητας. Και υπάρχουν χώρες, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κορέα, αλλά να μην γίνεται με τρόπο ασυντόνιστο αυτό. Ε, ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξέρετε το πρόγραμμα δράσης μας από τον Ιανουάριο και μετά, πέντε προτεραιότητες, 16 ειδικέ δράσεις και τώρα στο ιστορικό αυτό του προγράμματος σε πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως είναι η ε, αποστολή και παράδοση. Ε, θα προτείνουμε συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις. Ένα θέμα που είναι σημαντικό και για σας και για μένα είναι το πρόγραμμα δράσης για το λιανεμπόριο. Ε, κατόπιν ε, πρωτοβουλία της κυρίας Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Το Νοέμβριο του 2012 θα καταθέσουμε μία ανακοίνωση και θα υιοθετήσουμε την εγκάρση οριζόντια προσέγγιση της έκθεσης Κοράτσα Μπίλτ και θα ασχοληθούμε με τις εθνικές αποκλήσεις, με την πρόσβαση της ε, προσφοράς, ε, με τους καταναλωτές, με τον εφοδιασμό και θα λάβουμε υπόψη μας και το φόρουμ υψηλού επίπεδου για τον εφοδιασμό στα τρόφιμα για να δούμε ποιες είναι αθέμητες εμπορικές πρακτικές εκεί. Και τέλος, χωρίς να είναι το λιγότερο σημαντικό, ε, τα παίγνια στο διαδίκτυο. Δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ε, για τις υπηρεσίες. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που αφορούν την κοινωνία, όμως η προστασία των ανηλίκων, των νέων, καταπολέμηση ε, της εξάρτησης, ειλικρίνεια ε, των αγώνων ή των παιχνιδιών. Ε, χρειάζεται διοικητική συνεργασία. Υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη που ήδη συνεργάζονται μεταξύ τους. Ολοκληρώνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το μέλλον. Το μέλλον είναι πρώτα απ' όλα να υλοποιήσουμε τα όσα έχουμε αποφασίσει. 40 προτάσεις. Οι 12 από αυτές είναι η μοχλή για την πρώτη πράξη, τη μία εγκρίθηκε ήδη από εσάς. Υπάρχουν άλλες 30 από τις 50 που τις έχουμε ε, υλοποιήσει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε εκεί το συντομότερο να ολοκληρωθεί η πρώτη ενιαία πράξη, γιατί όλα αυτά τα μέσα ε, θα φέρουν ανάπτυξη, αλλά μέσω πρόθεσμα μόνο, γιατί χρειάζονται από 8 μέχρι 15 μήνες για να ε, γίνουν λειτουργικά, να εγκριθούν και να αρχίσουν να ισχύουν όλα αυτά. Λοιπόν, δεν αρκεί αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν ακόμα εμπλοκές, κατακαιρματισμοί που δεν έχουμε αντιμετωπίσει στην πρώτη πράξη για την ενή αγορά και γι' αυτό τώρα με 12 μοχλούς, προτάσεις κλειδιά για την ανάπτυξη που έχουμε εντοπίσει και προτείνει το Σεπτέμβριο, αφού ε, σας ακούσουμε και εσάς, θα φέρω 12 νέες προτάσεις. Αναφέρθηκα στο θέμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ένα άλλο θέμα με το συνάδελφο Άντορ, αλλά το λέω και με την επιφύλαξη της πρώτερης συμφωνίας του ε, κολεγίου, να υπάρχει δυνατότητα ε, μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, των συντάξεων στην Ένωση από μια χώρα σε ε, άλλη. Είναι ένα δεύτερο κύμα λοιπόν για την ενιαία αγορά και πάμε και προς την ψηφιακή ενιαία αγορά. 12 προτάσεις που θα έχουν αυτή τη ιδιότητα του μοχλού και θα φέρουν ανάπτυξη. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρε, προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένος. Ε, λοιπόν, σας ε, διανέμω τρία έγγραφα. Το πρώτο είναι, σας είπα, στα αγγλικά μόλις το έχουμε. Α, έχει ήδη διανεμηθεί, μαθαίνω, μάλιστα. Ε, είναι ενδιαφέρον αυτό το κείμενο. Καλύπτει όλες τις υπηρεσίες, και δείχνει ε, από ποια ευρωπαϊκά κείμενα ε, νομοθετικά καλύπτεται κάθε υπηρεσία. Ε, στη συνέχεια, το επικυροποιημένο ενημερωμένο πρόγραμμα εργασίας για το 12, τι έχουμε κάνει, τι μένει να γίνει και το τρίτο, επίσης ενδιαφέρον, η πρώτη πράξη για την ενιαία αγορά, οι 12 προτάσεις μοχλή, συν 50 συμπληρωματικέ. Ποιο επίτροπο είναι αρμόδιο για κάθε κείμενο και πού βρισκόμαστε. Ποιο έχει κάνει τι και τι απομένει να γίνει. Έτσι, ε, αυτά για να έχουμε όσο γίνεται ε, ένα μπούσουλα που θα σας οδηγήσει στη δουλειά σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τελειώνω εδώ. Well, thank you very much indeed. Uh, σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, για την όση συνήθω ευρύτατη και σαφέστατη ανακεφαλαίωση όλων των πρωτοβουλειών που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις λεπτομέρειες. Νομίζω πραγματικά καλό θα ήταν το Ευρωκοινοβούλιο για την πράξη της ενιαίας αγοράς να ετοιμάσει ένα ανάλογο κείμενο. Διότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ήταν χρήσιμο να είχε ένα τέτοιο εγγραφό όταν προσήλθε στο Συμβούλιο. Δεν το είχε, γιατί και εγώ βρέθηκα στη συνάντηση όπου συμφωνήθηκε να το υποβληθεί κάτι τέτοιο αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε και τις προσπάθειες για να γίνει αυτό. Η πρωτοβουλία να ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να αφοσιωθούμε σε αυτό είναι πολύ σημαντική για αυτή. Για μας. Διότι και η κοινοβουλευτική εργασία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πολύ καλύτερα. Ως τώρα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο κυριαρχείται από τις δημοσιονομικές και οικονομικές μέρημνες. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακούγονται και τα δικά μα τα σχόλια. Έχουμε χρόνο για συζήτηση. Απλώ θέλω να δω πόσοι συνάδελφοι θα ζητήσουν το λόγο. Ήδη Όλοι οι συντονιστές, θέλουν να παρέμβουν, οι αντιπρόεδροι. Μπορώ να δω ποιοι επίσης θα ήθελαν να προσθεθούν, η κυρία Βάιλερ, κάποιο άλλο. Μπορεί να το αποφασίσετε και αργότερα. Αλλά για να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ας ακούσουμε πρώτα τους αντιπρόεδρους μας και ας ακούμε ζεύγη ομιλητών. Η κυρία Πίτη Κάινεν και μετά η κυρία Βερνιό. Και θα ακούσουμε τους συντονιστές αντίστροφα, κύριο Ντεγιόν, κυρία Ρούλε, ο κύριος Μάντερς και η κυρία Γκέπχαρτ. Και μετά ο κύριος Σφάμπ. Σίγουρα και κάποιος ακόμη θα προσθεθεί. Ο κύριος Σφάμπ και η κυρία Βάιλερ. Μέχρι τώρα αυτούς το έχουμε στον κατάλογο αγορητών. Εάν κάποιος θέλει να προσθεθεί, με το Catch the Eye θα τα καταφέρουμε. Κυρία Πίτη Κάινεν, πρώτη αντιπρόεδρος, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, να συγχαρώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ για το αποτελεσματικό και αξιόλογο έργο που κάνει στην τομέα της ενιαίας αγοράς. Προσπαθείτε να συνδυάσετε τόσο διαφορετικές πτυχές όπως τη βιωσιμότητα, την κοινωνική διάσταση, το περιβάλλον, Καταρχήν, να πω κάτι που και ο Πρόεδρός μας το ανέφερε. Τον κατεπήγοντα χαρακτήρα που έχει η πράξη της ε, ενιαίας αγοράς και ε, τα όσα σχετίζονται με την ανάπτυξη στους δείκτες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά και οι δεσμευτικές πτυχές των διαπραγματεύσεων μαζί με την αποδοτικότητα των πόρων για το μέλλον. Ιδάλω δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τι υποχρεώσει μα. Ούτε να καλύπτουμε τι ανάγκε μα στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Επίση, να δείξω τρία ζητήματα για περαιτέρω σχόλια. Πρώτα απ' όλα, η απελευθέρωση των αγορών μα. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό με τρόπο σφαιρικό. Να ανοίξουμε διεθνώς και Επίσης και για δημόσιους διαγωνισμούς σε άλλες επίρους. Για την αποδοτικότητα των πόρων και τις καθαρές τεχνολογίες είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσο σκληρές ήταν διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το θέμα αυτό για την αποδοτικότητα της ενέργειας και την καθαρή τεχνολογία πρέπει να γίνουν προσπάθειες όχι μόνο εσωτερικώς για τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών αλλά και στο διεθνές επίπεδο τις εμπορικές μας σχέσεις και του δημόσιους διαγωνισμούς με άλλους εταίρους και με το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασία και περιβαλλοντική προστασία που απαιτείται. Χρειάζεται αυτό. Είναι κάτι που απαιτείται, αλλά Κάποιες από τις επιχειρήσεις ε, δεν ε, σέβονται τους κανόνες, ούτε θεωρούν ότι είναι επαρκή τα οικονομικά ωφέλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ίσοι όροι στον ανταγωνισμό. Επίσης, κάποια γρήγορα σχόλια. Για τα κεφάλαια κινδύνου υπάρχουν καινούργιες ιδέε πέρα από τον προτινόμενο κανονισμό. Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα κεφάλαια αυτά και να διευκολύνουν τη λειτουργία της ενία αγοράς. Και τέλος, θα ήθελα κάποια στοιχεία για την πρόταση που αφορά τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και τους κανόνες δικαίου εμπορίου. Διότι οι σχέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι σχέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες και τις πολυεθνικές είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερως. Ευχαριστούμε κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατά πρώτον να σας ε, συγχαρώ η εσωτερική αγορά αξίζει ιδέες καινοτόμε. Και εμείς λοιπόν πολλές φορές έχουμε ρίξει και ιδέες σε αυτή την Επιτροπή και το θεωρώ αυτό σημαντικό. Συγχαρητήρια κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχεστε συστηματικά για να συζητούμε αλλά το έχουμε δει και με τα θέματα που εξετάζουμε μαζί. Οι υπηρεσίε τη Επιτροπή οι ίδιε είναι πολύ ανοιχτέ στη συνεργασία μαζί μα. Κύριε Επίτροπε, σα συγχαίρω λοιπόν για αυτό που μόλι είπατε και που θυμήσατε αριθμού που αφορούν την εσωτερική αγορά. Διότι και εμεί, μάλλον οι συμπολίτε μα, βλέπουν πάντοτε την αγορά ω κάτι το τρομακτικό. Όταν όμω θυμίζει κανεί του αριθμού κατά αυτόν τον τρόπο, όπω κάνατε εσεί, το γεγονό ότι η ανάπτυξη που όλοι ευαγγελίζονται δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω τη εσωτερική αγορά. Σωστά λοιπόν δίνεται έμφαση όπω το κάνατε. Πρέπει σαφώ να επαναλαμβάνουμε ότι χρειαζόμαστε κοινωνική οικονομία. Κοινωνική. Η αγορά φτιάχνεται για τι επιχειρήσει, για το εμπόριο, αλλά και για του πολίτε. <clears throat> για κάποια από τα θέματα λοιπόν, ένα με ενδιαφέρει πρωτίστω, η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα ε, με μεγάλη χαρά σας άκουσα να λέτε ότι η ιδέα της επαγγελματική κάρτας είναι κάτι που το στήριξε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Ξέρουμε ότι αυτό το συζητούμε εδώ και πέντε χρόνια και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Η Μπάρμπαρα το ανέφερε προηγούμενο στο πηγαδάκι που είχαμε, κάποιες δυσκολίες με το Συμβούλιο, ακόμη και αν συζητούμε πολύ συχνά για το τι επίπεδο εναρμόνισης επιδιώκουμε, τι θα πρέπει να προσδοκούμε με την ε, όλη συζήτηση για αυτή την οδηγία. Εγώ θέλω να ευχηθώ να υπάρχει εναρμόνιση ως το δυνατόν πληρέστερη. Με σαφήνεια να υποδείξουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε και τις προάλλε το συζήτησα και στο δικό μας το κοινοβούλιο και στη Γερουσία με τους Γάλλους συναδέλφου, χωρίς παρόλα αυτά να πλήττουμε διαρκώ και να υποβιβάζουμε την αρχή της επικουρικότητας, ιδίως ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τις οικονομικές υπηρεσίες, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας. Θα μπορούσαμε νομίζω να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για τις κατεξουσιοδότης πράξης, για την μερική πρόσβαση και ούτω καθεξής. Όμως η όρη της συζήτησης μεταξύ μας είναι νομίζω θετική. Οι και οι σκιώδεις συζητητές ε, οργανώνουν συχνά συναντήσεις και με εμάς και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, είναι κάτι που μας επιβάλλεται για αυτές τη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν. Για την εσωτερική, την ενιαία μέλλον αγορά, ε, τονίσατε κάτι που νομίζω το βρίσκω και εγώ πολύ σημαντικό και άλλοι στην Επιτροπή μας. Το πρόβλημα της αμοιβαιότητας. Εδώ λοιπόν έχω μια ερώτηση. Στο κείμενο για τους δημόσιες προμήθειες διαγράφτηκαν δύο άρθρα για την αμοιβαιότητα επειδή υπήρχε νέα πρόταση κειμένου. Νομίζω καλό θα ήταν να επανεισαχθούν τα δύο αυτά άρθρα. Διότι υπάρχει εδώ νομίζω κενό, βεβαιό, ε, κενό νομικό και τα κείμενα δεν συμπίπτουν. Για τις ε, κορίσεις νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά ίσως να πετύχουμε τελικά μια συμβαστική λύση και για τις μελλοντικέ σα προτάσει για την μεταφορά συντάξεων και τα νέα εργαλεία για την καταπολέμηση των αθέμετων εμπορικών πρακτικών. Εδώ πραγματικά μπορείτε να υπολογίζετε και στη δική μα την βοήθεια. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε κάθε φορά δύο ερωτήσεις και να ακούσουμε συνέχεια τον Επίτροπο. Δεν θα καταφέρετε όλοι να θέσετε τρεις ερωτήσεις και παραπάνω. Το σημαντικό είναι να εστιαστούμε στα σημαντικά ζητήματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε στον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ την κυρία Κάινεν για τον τρόπο που εκτιμά το έργο μας. Όπως είπα και από την αρχή της θητείας μου, το ξέρουν και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών μου, ο κ. Κλάς που είναι εδώ, ο κ. Σάιμπερ, οι συνεργάτες μου από τη Γενική Διεύθυνση. Δεν είμαι ποτέ επίκης. Θέλω να είμαι πάντα άμεσος και επικοδομητικός και ενεργητικός της αποφασής μου για να μπορούμε να προχωρούμε και να γίνεται και δουλειά. Και να γίνεται δουλειά και γρήγορα. Η κυρία Πιτικάινεν παρατηρεί ότι όσα κάνουμε εγγράφεται στο... ναι, στην έκθεση Γκρέσπου που εγκρίνατε κι εσείς για την σφαιρική προσέγγιση. Αυτό είναι και η αξία της πράξης για την ενιαία αγορά, ότι διαρθρώνει μαζί σε ένα κείμενο πράγματα που ήταν χαμένα λίγο στο διάστημα μέχρι τώρα. Τα συνενώνει υπό τη λογική της κοινωνικής ε, οικονομίας, της ανταγωνιστικής αγοράς. <clears throat> Και οι τέσσερι όροι είναι πολύ σημαντικοί. Έχουν την ίδια σημασία η κοινωνική οικονομία τη ε, αγορά. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρήσει αυτό και μαζί με τον Όλυ Ρεν να υποβληθεί αυτή η πρόταση. Είναι μια σφαιρική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Δεν θέλουμε να ούτε στι κυρώσει να επιμείνουμε, ούτε στην παρακολούθηση, αλλά στην προώθηση ακριβώ τη ανάπτυξη. Εντοπίσατε του δείκτε, κυρία Πιτικάινεν. Τη σωστή χρήση των πόρων. Αλλά ιδίω του δείκτε τη ανταγωνιστικότητα. Κυρίε και κύριοι, εγώ είμαι πεπισμένο ότι είναι διπλή πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω προ την ανταγωνιστικότητα. Και ενδοκινοτικό, δηλαδή και ω προ τον υπόλοιπο κόσμο. Εντό τη κοινότητα θα πρέπει να υπάρχει benchmarking, δηλαδή γματοληψία, αλλά και σαφή απεικόνηση των αδυναμιών των επιμέρου χωρών. Κάθε χώρα έχει κάποια ατού, κάποια πλέον εκτήματα, η Ελλάδα όπω και οι υπόλοιποι, αλλά κάποιοι έχουν και δυναμίε. Μεγαλύτερε ή μικρότερε. Εάν λοιπόν γίνει μια πολύ πιστή απεικόνηση όλων αυτών των στοιχείων, θα γίνουν δημοσιονομικές προτάσεις, οικονομικές προτάσεις, σωστή χρήση των διευθυντικών ταμείων, με πολιτικές που θα ενισχύουν τα ισχυρά σημεία και θα αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες. Δεύτερη πρόκληση εξίσου σημαντική είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης να γίνεται αντιληπτή συνολικά ως προς τον υπόλοιπο κόσμο και τις περιοχές του. Για τις δημόσιες προμήθειες, όπως και στο κείμενο που ετοιμάζει ο κύριος Ταραμπελά, υπάρχει η ιδέα της ανάλυσης κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να ληφθούν υπόψη και αυτές οι πολυτομιακές, ή μάλλον οι ανησυχίες της αγοράς και των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, από όλους τους τομείς. Πρέπει να στηρίξουμε τα καινοτόμα στοιχεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τις δημόσιους διαγωνισμούς εκτός, τι εργαλείο διαθέτουμε. Υπάρχει διεθνής συνθήκη που ονομάζεται GP. E. Η συμφωνία για τις κυβερνητικές προμήθειες. Πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία. Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο, κυρία Πιτικάιναν, και πέρσι και προηγουμένω για να διαπραγματεύουμε το κείμενο αυτό με Αμερικανούς, με Ιάπωνες, Κορεάτες. Η Κίνα δεν έχει προσχωρήσει σε αυτήν την συνθήκη ακόμα, τη συμφωνία. Θέλουμε όμως μια ομαλότερη πρόσβαση στις αγορές τους γιατί κάποια στοιχεία είναι τελείως αποκλεισμένα. Ή κάποιες φορές οι Αμερικανοί φροντίζουν να προστατεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Ε, ε, οι Ιαπωνές έχουν διαφορετική αναλογία της αγοράς τους απελευθερωμένη σε σχέση με αυτό που έχουμε ανοίξει εμείς για εκείνους. Θα πρέπει λοιπόν να διακοπεί αυτή η τάση. Για αυτούς από εσά που ενδιαφέρει η ανοιχτή Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρεται στο πιάτο. Βέβαια και εγώ την απελευθέρωση θέλω, το άνοιγμα, τι ανταλλαγέ, τι εμπορικέ συναλλαγέ. Αλλά να μην είμαστε και αφελεί. Μπορεί να υπήρξαμε πριν 15-20 χρόνια, αλλά τώρα θα ζητήσουμε το άνοιγμα και των αγορών των άλλων. Άλλο όταν προβλέπεται αποκλεισμό ε, ε, από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Οι άλλοι τα χρησιμοποιούν ήδη. Οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνε ορισμένου κλάδου του αποκλείουν τελείω χάρη στην ε, συμφωνία αυτή. Κάποιε όμω ευρωπαϊκέ χώρε αυτό το κάνουν ατάκτω και χωρί καμία συνέπεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εδώ συνοχή στου διάφορου αποκλεισμού που ίσω επιβληθούν. Για τα κεφάλαια κινδύνου. Είναι μία από τι 12 προτάσει κλειδιά που συμπεριλαμβάνονται στην πράξη της ενιαίας αγοράς. Πρώτο μέρος. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει αν και το Κοινοβούλιο προχωρήσει αναλόγως και ελπίζω ότι θα έχουμε στο τέλος του χρόνου το διαβατήριο ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν τέτοια κεφάλαια κινδύνου να μπορούν να εργαστούν εύρυθμα στο επίπεδο και την κλίμακα της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει αυτό το νέο εργαλείο του Επιτήριου να συσχετιστεί με το πώς στηρίξαμε το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δηλαδή, το συζήτησα και με τον πρόεδρο της τράπεζας αυτής, να προσανατολίσουμε, να κατευθύνουμε ένα μέρος των κονδυλίων, των δανείων, που μπορεί να έχουν σκοπό τις επενδύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά να στηρίξουμε ουσιαστικά το κεφάλαιο κινδύνου και τις νέες, τις πρωτοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις. Κυρία Βερνιό, και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Για το κείμενο των επαγγελματικών προσόντων που τόσο πολύ έχετε δουλέψει, προχωρούμε παράλληλα. Είναι και για μένα προτεραιότητα να έχουμε μία βάση αμοιβές συνεννόησης για την κινητικότητα μεταξύ των διάφορων επαγγελματικών κλάδων στην Ευρώπη, ξεκινώντας από χαμηλά προς τα πάνω, διότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν αντιδράσεις επιφανειακές και συντηρητικές μάλιστα. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια εξάσκησης και εξοικείωσης. Η χώρα σας που είναι και δική μου, Βλέπουμε πώς αντέδρασε. Κίτρινη κάρτα έδειξε το κοινοβούλιο μας και ζήτησε επικουρικότητα. Ο κύριο Σαμπάτ μπορεί ίσω στα νέα του καθήκοντα να πείσει την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αλλά χάρη και στο δικό σα έργο και που εμεί παρακολουθούμε προσεκτικά, ίσω να εξηγήσουμε, να απαντήσουμε στι απορίε, να πούμε, γιατί δεν θέλουμε να ανατρέψουμε τα πάντα, οι ρυθμίσεις, τα κλειστά επαγγέλματα για αντικειμενικούς λόγους, συμβολιογράφοι και ούτω καθεξής, εκείνοι ε, παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να είμαι λοιπόν και εγώ ρεαλιστής. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Όμως με τον συνεχή διάλογο μπορούμε να αποδείξουμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία που αυτή η κάρτα κινητικότητα στην Ευρώπη θα μπορούσε να επιτρέψει να υπάρχει. Κυρία Βερνιό, για τα άρθρα 58-59 που όντως διαγράφησαν, Νομίζω ο κύριος Ταραμπέλα, ο εισηγητής σας, το γνωρίζει επαρκώς. Και βεβαίως και εγώ θα ήθελα η νομική ασφάλεια να ενισχυθεί. Εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία θα γίνει. Ε, ε, σας ευχαριστούμε. Τις ε, δύο επόμενες ερωτήσεις θα κάνουν ο κύριος Διόν και η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. τι προνομιακή μεταχείριση με την αντίστροφη σειρά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο και θα ήθελα να σας πω κάτι για τις εξελίξεις στη χώρα μου. Ξέρετε ότι στις 12 Σεπτεμβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές. Για πρώτη φορά στην ιστορία, εμείς το Σοσιαλιστικό Κόμμα ε, της Ολλανδίας έχουμε αγκαλιάσει την εσωτερική αγορά και θεωρούμε ότι φέρνει και ωφέλει και είναι συμβολικό αυτό πραγματικά. Ε, η εσωτερική αγορά ε, μπορεί να φέρνει καμιά φορά αρνητικές αντιδράσεις και αρνητικούς συνειρμούς, αλλά τελικά εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Γιατί τα λέω αυτά. Παραμένουν πολύ έντονες οι συζητήσεις για δύο πράγματα. Πρώτον, τα κοινωνικά δικαιώματα αφενός και αφετέρου ε, οι ίσοι κανόνες παιχνιδιού στην Ευρώπη. Δεν τους έχουμε δει πάρα πολύ να ισχύουν. Στην Επιτροπή μας εδώ για την εσωτερική αγορά είχαμε πολύ καλή συζήτηση και διμερός με τον Μάριο Μόντι, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Για τα κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να κάνουμε πρόοδους, αλλά και στα δημοσιονομικά πρέπει να κάνουμε πρόοδους. Και για να είμαι ειλικρινής, ε, Ε, δεν έχουμε δει πολλά πράγματα εκεί με εξαίρεση την οδηγία για τις υπηρεσίε. Τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, τα κοινωνικά δικαιώματα να γίνουν σεβαστά και να ορίζονται κιόλας. Αλλιώς θα υπάρχει πάντα ένα τμήμα της κοινωνίας και ορισμένοι μιλούν για τη μισή κοινωνία που θα είναι εκτός και θα ε, παραμένει κατά της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό και εγώ ε, ζητώ παρακαλώ να κοιτάξουμε και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ας πούμε, ίσως μισθός για ίσης αξίες εργασίας και ε, προστασία του δικαιώματος της απεργίας. Σε ό,τι αφορά τους ίσους κανόνες παιχνιδιού και τα δημοσιονομικά, για το φόρο Επί των κερδών της επιχείρησης ε, δεν θα πρέπει να είναι σε θελοντική βάση. Έχει έρθει η ώρα να ρυθμιστεί αυτό στην Ευρώπη, να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο και εκεί δεν βλέπω και φιλοδοξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνει πρόοδος. Αυτό είναι το δεύτερο. Λοιπόν, αν ρυθμίσετε αυτά τα δύο, κοινωνικά δικαιώματα και ε, ε, ένα ελάχιστο φόρο επί των κερδών των επιχειρήσεων, θα προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούω πολλές ε, αντιδράσεις από επιχειρήσεις ε, ε, καταργείτε κάποιους κανόνες, καλό είναι αυτό, ε, για να μειώσετε τη γραφειοκρατία, αλλά μετά φέρνετε νέους κανόνες και οι επιχειρήσεις λένε ότι τελικά επιβαρύνονται περισσότερο. πρόσβαση στη χρηματοδότηση επίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα θέμα και πρόβλημα. Δηλαδή, μου ζητούν αντί ε, πρόγραμμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, καλό θα ήταν ε, σε επιμέρους προγράμματα όπως είναι το ερευνητικό πρόγραμμα το Horizon να υπάρχει ένα κεφάλαιο εκεί ειδική πρόνοια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θεωρούν πιο σκόπιμο αυτό. Και ένα τελευταίο για την εγκληματικότητα. για τις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιθετική εξαγορά και στις απάτες που γίνονται εκεί απέναντί τους. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόν και κύριε Ριουλέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που έρχεστε πάντα εδώ στις συζητήσεις μας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις καλές προτάσεις περσινές και την πράξη για την ενιαία αγορά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες καθόλου. Θα ήθελα να εκφράσω μία παράκληση. Και αυτό αφορά το ζήτημα των αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων. Είναι 20% του ΑΕΠ και η νομοθεσία είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Εγώ τα έχω διαβάσει λίγο γιατί κάνω και τροπολογίες σχετικά. Αλλά δεν μπορώ πάνω να πω ότι ακόμα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιέζεται χρονικά και αυτό φαίνεται από το κείμενο. Έχει ελλείψεις λόγω της χρονικής πίεσης. Λοιπόν, μην μας πιέσετε ε, παρακαλώ να μας αφήσετε λίγο χρόνο να δούμε με την ησυχία μας ήρεμα ε, τι θα κάνουμε, πώς θα έρθει μια καλή και σωστή νομοθεσία για να είναι πραγματική ελάφρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τους Δήμους και τις κοινότητες. Στα γερμανικά λέμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και ε, πραγματικά χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Ένα άλλο που θέλω να φέρω είναι ακριβώς με τις δημόσιες συμβάσεις πάλι για την αμοιβαιότητα. Εκεί έχω μεγάλες επιφυλάξεις Θεωρώ πραγματικά ότι και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σε βάθος. Δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι εμείς στην Επιτροπή μας, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε οπωσδήποτε. Αν θέλουμε να επιβάλλουμε την αμοιβαιότητα, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς, ας πούμε τα κομπιούτερ, που είναι υποχρεωτικό να απευθυνόμαστε σε τρίτες χώρες. ICT, τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Προσοχή όταν μιλούμε για μέσα αμοιβαιότητας να μην ε, ακροτηριαζόμαστε από μόνοι μας σε κάποιους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Να μην είναι πάρα πολύ σκληρά και άκαμπτα αυτά τα μέτρα. Και μια τελευταία ερώτηση. Με ενδιαφέρον διάβασα το νέο σας πρόγραμμα και το θέμα της διακυβέρνησης και όλα αυτά και πολλά τα υποστηρίζω και τα βρίσκω ωραία και σωστά. Αλλά έχω μια ερώτηση ισχύει αυτό που λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις αδυναμίες και ε, τα ισχυρά σημεία των κρατών και να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες. Κάτι άλλο που λέτε συχνά ε, στα έγγραφα είναι οι υπηρεσίες της οικοδομικές ε, ε, δραστηριότητες, στο κατασκευαστικό τομέα και αγωνιούν πολλά κράτη-μέλη. Τι εννοείται ακριβώς εκεί να ανοίξει η οδηγία και η αγορά. Μπορεί να υπάρχουν επαγγέλματα που θα πρέπει να ε, σπάσουν κάποιες ρυθμίσεις, είναι κλειστά, αλλά υπάρχουν και επαγγέλματα που συνδέονται με την ασφάλεια. Κοιτάξτε τι γίνεται ας πούμε με κάποιους που κάνουν εγκαταστάσεις υγραερίου ή ενέργειας Οπότε αν την απορριθμίσουμε τελείως στην αγορά μπορεί να υπάρχει και θέμα ασφάλειας στα τεχνικά αυτά επαγγέλματα. Και για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι κάτι που χρειάζεται προσοχή και τα ισχυρά και τα δύναμα σημεία. Σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουν και ισχυρά και η δικιά μου χώρα και όχι μόνο η δικιά μου, έχει μια μορφή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που είναι διτή, παράλληλη, σχολείο και άσκηση. Και εκεί είναι μικρότερη η ανεργία των νέων από ό,τι σε άλλε χώρε. Λοιπόν, αυτά τα ισχυρά να τα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και να μην τα αποδυναμώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος. Να απαντήσω καταρχάς στον κύριο Ντεγιόγκα. Δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει στο πολιτικό του κόμμα προκειμένου να γίνει αυτή ε, η ε, προσέγγιση με τις ευρωπαϊκές αυτές πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρθηκε, προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη χώρα του και θα αποτελέσει θετικό παράδειγμα πιστεύω και σε άλλες χώρες όπου δεν έχουμε απαραίτητα τις ίδιες εξελίξεις. Ε. Δεν αναφέρομαι σε κάποια χώρα. Πάντως πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό και το λέω πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ιδεολογική προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενιαία αγορά αποτελεί το δικό μας ενιαίο κοινό χώρο για την οικονομική και την κοινωνική ζωή. Και αυτό που έλεγα στου Έλληνε λίγε μέρε πριν τι εκλογέ και στον πληθυσμό τη Ιρλανδίας είναι ότι συνειδητοποιώ ότι καταβάλουν πολύ σημαντικέ προσπάθειε έχουν κάνει πάρα πολλέ θυσίε, πάρα πολλέ φορέ είναι εξοργισμένοι. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι στον σημερινό κόσμο, και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν άλλωστε και εκλογή σα. Αν ανοίξουμε τα μάτια και δούμε ξεκάθαρα τα πράγματα, βλέπουμε ότι η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βραζιλία, πώ αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τον κόσμο οι χώρε αυτέ και πώ μπορούμε εμεί μέσα από τον κόσμο να προασπίσουμε τα συμφέροντά μα και τι αξίε μα. Δρώντα ω μεμονωμένε χώρε, ω Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα ή όλοι μαζί συλλογικά. Νομίζω ότι κάθε ψηφοφόρο θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα αυτό για τον ίδιο και για τους άλλους. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μας ακούσουν περισσότερο, προκειμένου να καταφέρουμε να πείσουμε τους εταίρους μας περισσότερο. Σαφώς μπορούμε να είμαστε πατριώτες, σαφώς μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας, αλλά παράλληλα πρέπει και οφείλουμε να είμαστε και Ευρωπαίοι. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα καθίστανται πολύ πιο δύσκολα, αν δρούμε απλώς για το δικό μας συμφέρον περιχαρακωμένοι στη χώρα μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα αυτό και υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο ακόμα προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την ευκταία αυτή πρόοδο. Να μειώσουμε για παράδειγμα τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία δεν υπάρχει μόνο στις Βρυξέλλες. Σίγουρα υπάρχει και στις Βρυξέλλες, αλλά γραφειοκρατία εμφανίζεται και αλλού. Θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα κάποια κοινωνικά δικαιώματα και προς αυτό Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Άντρες, ο συναδελφός μου, έκανε μια πρόταση όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζομένους. Στα πλαίσια του πακέτου του αποκαλούμενου Μόντι 2, Κάναμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα κοινωνικά συλλογικά δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες. Εμείς αναλάβαμε τις ευθύνες μας σε σχέση με την πρόταση αυτή και θα ξεκινήσουν τώρα οι συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο παράλληλα. Κύριε Ντεγιόνγκ, πρόσεξα ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε για τη φορολογία. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο προποθέσει προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο στη φορολογία στα πλαίσια τη ενιαία αγορά. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει πρωτοβουλίε. Και δεύτερον, το Συμβούλιο πρέπει και αυτό, με τη σειρά του, να αλλάξει συμπεριφορά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Γιατί στον τομέα αυτό τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς ομοφωνία. Εκτός και αν χρησιμοποιηθεί μια διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπει την ενισχυμένη συνεργασία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει την πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σωστά την δουλειά της. Ο συναδελφός μου Σεμέτας είναι ένας πολύ θαραλέος επίτροπος γιατί το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και μέσα σε δύο χρόνια έκανε τρεις συγκεκριμένε προτάσεις εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες εγώ υποστήριξα όσον αφορά την οικολογική φορολογία, όσον αφορά τον φόρο για τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές, το οποίο θα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα, καθώς επίσης και την κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείες επιχειρήσεις. Δεν αναφέρομαι σε φορολογικό στελεστή, αναφέρομαι σε φορολογική βάση. Το υπάρχει δηλαδή ένα ελάχιστο επίπεδο όσον αφορά την φορολογία των εσόδων των κερδών. Στα πλαίσια λοιπόν μιας ενίας αγοράς 27 κρατών μελών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία συμφωνία και αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία τουλάχιστον να υπάρχει μία ενισχυμένη συνεργασία και αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μία κοινή φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις αυτό θα αποτελέσει πραγματική πρόοδο. Καταγράφω πάντως τις προτάσεις που κάνετε σε σχέση με αυτό και ειλικρινά πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό έχει πραγματικά σημειώσει πρόοδο και έχει δείξει ότι έχει φιλόδοξες προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε επίσης και στη γενικότερη αναθεώρηση και επικαιροποίηση του φόρου τη προς θέμενης αξίας. Κύριε Τεγιόνγκ, συμφωνώ επίσης με τις απόψεις όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Προεδρός σας, ο κύριος Χάρμπορ, με την συνεργασία επίσης του Επιτρόπου κύριου Ταγιάννη, εργάζεται και αυτός προκειμένου να έχουμε αυτή την ε, αποκαλούμενη ε, σύμβαση Ευρώπη μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να καταφέρουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας μάλιστα και ένα δίκτυο των εμπορικών επιμελητηρίων των κρατών μελών. Πήγα στη Γερμανία και είδα πραγματικά ότι το εκεί δίκτυο είναι πάρα πολύ επαγγελματικό, έχει πολύ υψηλή ποιότητα. Επίσης αυτό που είδα είναι ότι στη Γερμανία γίνεται κάθε χρόνο μία έρευνα σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις όσον αφορά την απτυξή τους, τα αποθέματά τους, τις οικονομικές προβλέψεις. Κατά αυτόν τον τρόπο ένα χρόνο από τον προτέρων, χώρες όπως η Γερμανία είναι σε θέση να έχουν πολύ ακριβείς οικονομικές προβλέψεις όσον αφορά τι επιδόσεις των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ εμπορικών επιμελητηρίων προκειμένου να διαχέονται τέτοια έγγραφα τα οποία θα μας βοηθούν να πούμε ότι κοιτάξτε ε, το Small Business Act, η ε, ενιαία αγορά γενικότερα, οι δημόσιες συμβάσεις, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες για τις επιχειρήσεις αυτές. Να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για όλα αυτά τα ζητήματα. Και ξέρετε, ως προς τη δανειοδότηση κάναμε κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις και μέσω της ε, Συμφωνία τη Βασιλεία. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι, και τουλάχιστον σε όλε τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει που υπάρχουν για τι τράπεζε, να μην ζημιωθούν σε καμία περίπτωση οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δανειοδότηση και να υπάρχουν και απαραίτητε εγγύησεις προκειμένου να υλοποιείται στην πράξη η δανειοδότηση αυτή. Με τον κύριο Ταγιάννη λοιπόν πρόκειται να συντάξουμε το έγγραφο αυτό το οποίο θα πάει άμεσα σε όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, εγγράφο και μέσω διαδικτύου ενδεχομένω. Όσον αφορά τώρα τις ε, εκχωρήσεις, τις παραχωρήσεις, ε, με τον κύριο Ζουβά θα προσπαθήσω να δω, τον εισηγητή σας δηλαδή, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον ε, διοικητική πίεση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νομική ασφάλεια για τις μικρομισές επιχειρήσεις όσον αφορά τις ε, εκχωρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφανές νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις εκχωρήσεις υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τις δραστηριότητες αυτές. Θα εξετάσω πάντως περισσότερο να δω για ποιο λόγο έχετε την ανησυχία αυτή, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι προτάσεις μας προσθέτουν περισσότερη γραφειοκρατία. Κυρία Ρούλε, όντως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 18-20% του ΑΕΠ θα πρέπει σαφώς να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες αυτές που έχουμε για να δημιουργήσουμε μια οικονομική ανάπτυξη και για να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τελικά καλύτερα τις δημόσιες αυτές συμβάσεις που θα μπορούσαν να προωθήσουν και τα κοινωνικά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινοτομία. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα και το πόσο πιεστικό είναι, οι δημόσιε συμβάσει αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τομέα και μια βασική εμπλοκή είναι βασικά η γραφειοκρατία. Το διοικητικό αυτό άκτο το οποίο έχουμε πει ότι θέλουμε να μειώσουμε δραστικά. Και αυτό ισχύει βέβαια και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εύχομαι πραγματικά να προχωρήσουμε γρήγορα και αυτό επιθυμούν άλλωστε και οι αρμόδιοι υπουργοί και έχω παρατηρήσει πολλέ φορέ άλλωστε και το, ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ καλά και πολύ γρήγορα και ελπίζω ότι αυτό θα κάνει και για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Όσον αφορά την αμοιβαιότητα τώρα, Κυρία Ρούλε, για άλλη μια φορά θέσαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις. Εξήγησε ήδη δύο φορές για ποιο λόγο χρειαζόμαστε το μέσο αυτό της ε, αμοιβαιότητας. Δύο επιτροπέ ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Ελπίζω να καταφέρουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και ο κύριο Δεγκούτ και εγώ χρειαζόμαστε πραγματικά να έχουμε την αμοιβαιότητα. Ο κύριο Δεγκούτ για να ανοίξουν οι αγορέ και εγώ χρειάζομαι την αμοιβαιότητα προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία εφαρμογή του GPA, τη Συμφωνία Περιδημοσίων Συμβάσεων στην Ευρώπη καταλαβαίνετε ότι ε, σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να δούμε αν μπορεί από τη μία πλευρά στις δημόσιες συμβάσεις να χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό, αλλά θα πρέπει από την άλλη πλευρά επίσης να δούμε αν ε, το μέσο αυτό στο επίπεδο 1 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Σε 30 περιπτώσεις ετησίως έχουμε δει. Και έχουμε επίσης και την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε φορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα ελέγχει πώς εφαρμόζεται η αμοιβαιότητα και θα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η προβλεπόμενη διαδικασία να τυχαίνει κατάχρηση. Όσον αφορά τώρα τον κατασκευαστικό κλάδο και τις σχετικές υπηρεσίες, η οδηγία για τις υπηρεσίες καλύπτει και τον κλάδο αυτό Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ανοίξουμε πάλι την οδηγία αυτή, πάντως σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επιμείνετε προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, πιστά και ένα από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στο κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την απασχόληση, είναι ότι πολλές φορές εμφανίζονται προβλήματα ανάμεσα στην οδηγία για τις υπηρεσίες και κάποιες άλλες οδηγίες, όπως για παράδειγμα αυτή για τα επαγγελματικά προσόντα, ή ενδεχομένως και κάποια άλλα νομοθετικά κείμενα. Θα πρέπει ακριβώ να δούμε λοιπόν πού εντοπίζονται τα προβλήματα, πού έχουμε μπλοκές και πού υπάρχουν αντιφάσει ανάμεσα στα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, τα οποία διευθετούν την ενιαία αγορά. Κάτι αντίστοιχο κάναμε και στον τομέα του τουρισμού. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δούμε και εκεί πώς λειτουργούσαν τα πράγματα, γιατί και ο τουρισμός εντάσσεται στην οδηγία και τις υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρόκειται να βάλουμε κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά προσόντα τώρα ξέρω ποια είναι τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη χώρα σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να θέσουμε ένα αμφιβόλο το εναλλακτικό σύστημα κατάρτισης το οποίο υπάρχει σε χώρες όπως η Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες το σύστημα αυτό πραγματικά καταρτίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και επαγγελματίε όπως οι νοσοκόμοι. Πρόκειται για ένα σύστημα διπλής κατάρτισης. Το περιγράψετε και εσείς, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα. και επιτρέπει να κρατάμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο την ενέργεια των νέων στη Γερμανία. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό. Δεν θα ήθελα να ευνοήσω τα opting-out. Θα πρέπει πάντως να βρεθεί μια επικοδομητική λύση προκειμένου να καταφέρουμε να διατηρήσουμε όλα αυτά τα οποία λειτουργούν σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα απλώς να επιβάλλω αυτά τα οποία α, λέω ή λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε ότι αποφασίσουμε κοινοτικά με κάποια πολύ θετικά εθνικά παραδείγματα όπως αυτά της Γερμανίας. Um, Έχουμε 20 λεπτά μόνο, οπότε πρέπει να είστε πολύ σύντομοι στι ερωτήσει σα. Προσθέθηκε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κάποιο άλλο έχει ζητήσει το λόγο επιπλέον. Ωραία. Α ακούσουμε τον κύριο Μάντερ και την κυρία Γκέπχαρτ πρώτα. Δύο επόμενε ερωτήσει. Μετά κύριο Σφαμπ, κυρία Βάιλερ και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. 20 λεπτά, 10 λεπτά για κάθε γύρο προκειμένου να προλάβουμε και τι τελευταίε ερωτήσει. Δεν είναι ότι θέλω να πιέσω τον Επίτροπο. Κύριε Μάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπω εδώ και υποστηρίζουμε αυτά που μας παρουσιάζετε. Η κρίση και η έξοδος από την κρίση έχει μία απάντηση, μια ε, καλώς λειτουργούσα νεα αγορά, καλές οι οικονομίες και καλές οι ε, περικοπές, αλλά ακόμα καλύτερη πραγματική οικονομία. Μιλήσατε για την απλούστευση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Στον ΠΟΕ θα αυξήσετε τα κατόφια τις κατώτατες τιμές. Γι' αυτό θα ήταν μεγάλη απλούστευση. Γιατί νομικά ως Κοινοβούλιο εμείς δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Έχω την ε, αίσθηση ότι οι καινοτομίες ε, μπορούν να ενισχύονται από τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή μικρομεσές επιχειρήσεις ε, επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα και μπορούν έτσι να τα κάνουν γνωστά στις δημόσιες αρχές και στην αγορά. Επίσης, ε, σήμερα η παραποίηση προϊόντων είναι μάστιγα ε, αξίας ε, ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ έχουμε παραποιημένα προϊόντα, ευρωπαϊκές μάρκες, σήματα, παράγονται στην Κίνα και πολλούνται ανά τον κόσμο. Ξέρω ότι ο κύριος Ντεχούχτ χτες έκανε μια προσφυγή, ε, δεν ξέρω τι θα βγει. Ε, επηρεάζει την ευρωπαϊκή οικονομία, την απασχόληση. δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, όπως δεν ξέρουμε και το αποτέλεσμα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κατά τα άλλα. Ε, επίσης, ε, είπατε ότι θέλετε να έρθει ένα δίκαιο για τα διπλώματα τεχνίας και αυτό το καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Μόνο το Άμστερνταμ δεν ζήτησε το δικαστήριο <laughs> περίπου ε, από όλες τις πόλεις που ερίζουν για την έδρα του. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Και ελπίζω πάρα πολύ αυτό το θέμα της έδρας να μην μπλοκάρει το όλο ζήτημα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και ε, θα ήταν μεγάλη βοήθεια ακριβώς για μικρές, μισές επιχειρήσεις καινοτόμε και υγιείς. Έχει έρθει η ώρα επιτέλους να ληφθεί η απόφαση γι' αυτό και ελπίζω να γίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τον τρόπο με τον οποίο μας αναφέρετε πάντα με μεγάλη ειλικρίνεια ε, τα πεπραγμένα σας, τις προθέσεις σας και τα συζητάτε μαζί μας. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη γενικότερη αρχή ε, που θεωρώ πολύ καλή, ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση και προσέγγιση ε, να λαμβάνουμε υπόψη πάντα όλους τους τομείς πολιτικής. Και τώρα επανειλημμένα αναφερθήκατε στην οδηγία των υπηρεσιών που είναι πάρα πολύ σημαντική ιδιαίτερα στην εφαρμογή της. Και δεν μπορώ παρά να σας υποστηρίξω και ως πρώην εισηγήτρια χρειάστηκε πολύ κόπος για να περάσει αυτό το κείμενο και τώρα θέλουμε και ως βουλευτές βεβαίως να υλοποιείται σωστά. Στην οδηγία όμως για τις υπηρεσίες και στο πρώτο άρθρο ε, υπάρχει μια πολύ σημαντική διάταξη που συμπεριλάβαμε και αυτή ονομάζεται κοινωνική ρήτρα. Δηλαδή τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και το εργατικό ή τα δικαιώματα απεργίας ας πούμε, δεν θα πρέπει να διακυβεύονται ή να αμφισβητούνται από την εφαρμογή της οδηγίας. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η συνάδελφος Μπενατέτ Βερνιού προηγουμένως. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, στο μεταξύ έχουμε και την υποχρέωση ε, οι οικονομίες να είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και να λαμβάνει υπόψη αυτό το κοινωνικό, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, θα πρέπει αυτό να κυριαρχήσει περισσότερο στην πολιτική. Και έχω πάντα την εντύπωση ότι όχι εσείς προσωπικά, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κολέγιο των Επιτρόπων, παραμένει πάρα πολύ επιφυλακτικός και διστακτικός σε αυτά τα θέματα. Και σας ερωτώ, εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να φροντίσουμε η κοινωνική ρήτρα που είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε οι πολίτες μας να δεχθούν την εσωτερική αγορά και να διαλυθεί αυτός ο σκεπτικισμός και να ε, ξαναδοθεί στην Ευρώπη μια θετική προοπτική. Να βλέπει ο κόσμος δηλαδή ότι είναι ε, μια υπόθεση για το μέλλον του. Αυτό πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε να το προωθήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντερς γιατί μα συμμεθύμισε και αυτό ότι η ενιαία αγορά, ότι δεν αποτελεί τη μόνη απόντηση στην ε, πρόκληση της οικονομική ανάπτυξη, αποτελεί ενδεχομένω την πρώτη απάντηση που θα πρέπει να δώσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση. Η ενιαία αγορά λοιπόν αποτελεί την βάση, την πλατφόρμα για την οικονομία αν κατακαιρματιστεί η βάση αυτή σε 27 επιμέρους εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τη φορολογία για παράδειγμα ή την ε, διοίκηση ή αν δημιουργηθούν 27 διαφορετικές συνθήκες γραφειοκρατίας, τότε δεν μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε και δεν θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε ούτε τις δημόσιες ούτε τις α, ε, α, ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και μία πολιτική πλατφόρμα και με ορισμένους συναδέλφους μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργαζόμαστε μια ιδέα που δεν έχει γίνει απόλυτα κατνοητή, μια νέα βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη, να καταφέρουμε να ξαναβρούμε μια ικανότητα βιομηχανικής παραγωγής, έτσι ώστε να μην είμαστε μόνο στην Ευρώπη ένας χώρος όπου καταναλώνουμε κινέζικα προϊόντα ή στην καλύτερη περίπτωση δρούμος υπεργολάβη για την βιομηχανική παραγωγή άλλων είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βρούμε μια νέα πολιτική που θα καταφέρει να συνοδεύσει την πολιτική των εθνικών ενισχύσεων που δίνονται για τις, ε, τη βιομηχανική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σταθερή κοινή βάση όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Το κατόφλι των δημόσιων συμβάσεων στο οποίο αναφερθήκατε κύριε Μάντερς αποσαφηνίζεται κυρίως στα πλαίσια του GPA. Πρόκειται για μια πολυμερή διεθνή συμφωνία, στα πλαίσια της οποίας έχουμε θέσει συγκεκριμένα όρια. Είναι επομένω πολύ δύσκολο να επαναχωρήσουμε αυτή τη στιγμή. και ουσιαστικά προσπαθήσαμε σε σχέση με το GPA να προσαρμόσουμε πολλέ από τι συμφωνίε που έχουμε με τρίτε χώρε. Όπου όμω είναι δυνατό αυτό το κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, αυτό γίνεται και στην πρόταση που σα παρουσίασα για τι κοινωνικέ υπηρεσίε και τι σχετικέ δημόσιε συμβάσει. Καταφέραμε να αυξήσουμε τα όρια τα οποία προβλέπουμε εκεί, προκειμένου να διευκολύνουμε την ε, παροχή των ε, υπηρεσιών αυτών μέσω δημοσίων ε, συμβάσεων. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το ότι έχουμε ακριβώς το κατόφλι αυτό, τα όρια αυτά είναι πολύ, σημαντικά, πολύ σημαντικό για την ενιαία αγορά. Γιατί αν αυξήσουμε πάρα πολύ το κατόφλι, τότε αυτόματα θα μπορούσαμε να μειώσουμε τελικά και τις εγγύσεις για ζητήματα διαφάνειας και πρόσβασης της αγορά, στην αγορά για ορισμένες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια όμως της συζήτησης που κάνουμε βάσει της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η όλη συζήτηση για το κατόφλι αυτό να ανοιχτή αρκεί να μην πειράξουμε τα όρια τα οποία έχουμε θέσει διεθνώς στα πλαίσια του GPA. Όσον αφορά την παραποίηση, συμφωνώ απόλυτα μαζί, με τη δική σας την ανάλυση. Και εγώ με, τον συναδελφό μου, με τους συναδέλφους μου, τα Γιάννη και Σεμέτα, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την καθημερινή αυτή καταπολέμηση της παραχάραξης, της παραποίησης. 200.000 θέσει εργασία κάθε χρόνο χάνονται εξαιτία τη παραποίηση, αλλά και απειλείται επίση η δημόσια υγεία μέσω τη παραποίηση φαρμάκων, για παράδειγμα. Και απειλούνται κυρίω οι πολίτε από τι πιο φτωχέ χώρε, Για παράδειγμα, στην Αφρική υπάρχουν πάρα πολλά παραποιημένα φάρμακα τα οποία φτάνουν τελικά στην Ευρώπη μέσω των δικών μας τολιμένων μάλλον με συγχωρείτε, πολλά παραπημένα φάρμακα μέσω των δικών μας λιμένων φτάνουν σε χώρες όπως η Αφρική και αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά παράδεκτο. Η πρώτη απάντηση που έχουμε για την παραποίηση είναι καταρχάς να υπάρχει η σωστή προστασία των εφευρέσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μέσω εμπορικών ονομασιών. Θα αναφερθώ και σε αυτό λίγο αργότερα. Και επίσης πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σύνορα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, που διαθέτει και η υπηρεσία του Αλικάντε, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη κατάρτιση, μια συστηματική κατάρτιση για όλες τις δημόσιες αυτές υπηρεσίες που λειτουργούν μεθοριακά και θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων αυτών, καθώς επίσης και απαραίτητη πυρογνωμοσύνη για να καταφέρουμε να εντοπίζουμε τα παραποιημένα προϊόντα. Θα πρέπει επίση με το γραφείο του Αλικάντε να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε και ιδίω οι νέοι πόσο στοιχίζει τελικά η παραχάραξη, η παραποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη διαπαιδαγώγηση σε σχέση με αυτό. Και τέλο, θα πρέπει επίση να συνεργαστούμε και με τι χώρε αυτέ από τι οποίε έρχονται παραποιημένα, παραχαγμένα προϊόντα. Και έχω έρθει σε επαφή με την Αφρικανική Ένωση πολλέ φορέ. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία που έχουμε με την Αφρικανική Ένωση. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε μια task force όπου συζητάμε συγκεκριμένα ζητήματα όπως η παραποίηση και έχουμε βέβαια και χώρες όπως η Κίνα που σιγά σιγά αρχίζει και συνειδητοποιεί πόσο σημαντική είναι η πρόκληση αυτή. Όσον αφορά τώρα τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, τα οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκέπχαρ, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω τώρα σε αυτό, είναι το τελευταίο πρόβλημα βέβαια που θα μπορούσα να είχα φανταστεί. Έχουμε επιλύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που είχα ποτέ φανταστεί θα μπορούσαν να προκύψουν. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα προέκυπτε μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου ένα πρόβλημα, μια όσον αφορά τα 47 άτομα τα οποία θα εργαστούν στο γραφείο αυτό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πιο σημαντική είναι η πρωτοβουλία αυτή και θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να συμφωνήσουν για την κατάρτιση του γραφείου αυτού και ελπίζω ότι θα σημειωθεί κάποια πρόοδος και την επόμενη εβδομάδα. Από όσο γνωρίζω, κάποιοι Ολλανδοί υπουργοί είχαν κάνει και αυτοί κάποιες προτάσεις. Δεν ξέρω όμως αν θα διευκολυνθούν πάρα πολύ τα πράγματα να εμφανιστεί τώρα και μια τέταρτη πόλη υποψήφια για την έδρα του οργανισμού αυτού. Κύριε Γκέπχαρτ, πολύ σύντομα θα ήθελα να αφαιρθώ στη δική σας την παρατήρηση που ήταν πολύ συγκεκριμένη. Πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση της ενίας αγοράς. Αυτό μας βοηθά, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ε, συναδέλφους μου να καταφέρουν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια της σφαιρικής ατζέντα για την νέα αγορά που πρώτη φορά παρουσιάσαμε. Είναι πολύ καλύτερο να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο με έναν τρόπο καθαρά συλλογικό από το να λειτουργεί ο κάθε επίτροπος στον τομέα του ξεχωριστά. Και βέβαια και εγώ και άλλοι Επίτροποι, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες και ξέρετε επίσης ότι θέλω να υπάρχει μια ισορροπία στα πλαίσια της πράξης για την ενιαία αγορά κάθε φορά που αναφερόμαστε σε πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία αυτή με τους 12 μοχλούς. Ένας από τους μοχλούς ήταν η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίες οι προτάσεις αυτές. Στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα, αναφερόμαστε σε 3-4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι επικερδείς. Η γραμμή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλωστε κυρίως ο πρόεδρος Μπαρόσο το έχει πει και υποστηρίζει τη γραμμή αυτή. Η γραμμή μας λοιπόν έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την άκαμπτη γραμμή της απόλυτης ε, απορρίθμιση απελευθέρωσης τη αγορά την οποία είχαμε πριν από κάποια χρόνια. Έχουμε ε, προχωρήσει από το στάδιο αυτό, έχει εξελιχθεί η στάση μα και προφανώ αυτό έχει συμβάλει και η οικονομική κρίση. Now, the last... Και τώρα, τρεις τελευταίοι ομιλητές για το πρωί, ο κ. Φαμπ, η κυρία Βάιλερ και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Όσο δυνατόν συντομότερα για να τελειώσουμε καιρός. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτά που μόλις είπε ο, ο Μισελ Μπαρνιέ, αυτά που είπε τώρα κύριε Επίτροπε, είναι ε, και θέμα επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα ε, άκρος ε, φιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σήμερα και το ίδιο με την ανάπτυξη. Είναι θέμα επικοινωνίας. Από τη στρατηγική της Λισαβόνας από το 2001 συζητάμε για ανάπτυξη και στρατηγικές κάναμε που δεν ε, απέδωσαν. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς επικοινωνούμε αυτά που θέλουμε για να έχουμε και το αποτέλεσμα. Γενικά για την πράξη για την ενιαία ώρα, το είπε και η κυρία Ρούλε είναι πάρα πολύ θετικό που βλέπουμε πόσο ασχολείται ο Επίτροπος να έχουμε κανόνες ενιαίους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από συνεννόηση είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που κάνετε με τις άλλες γενικές διευθύνσεις ε, και είναι πάρα πολύ θετικό και ελπίζω να αξιολογείτε και μια δουλειά ουσίας που χρειάζεται επιμονή και διάρκεια. Είναι σημαντικό οι οδηγίες να όλες να είναι οριζόντιες εγκάρσεις, να έχουν συμφωνήσει οι υπηρεσίες και οι πολιτικές. Τελικά όμως οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλα. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα. Και έρχομαι στην πρόταση για την καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά. Η κυρία Γκέπχαρτ το είπε επίση. Η οδηγία για τι υπηρεσίε μετά από λίγα χρόνια τη θέση σε ισχύ για πρώτη φορά αξιολογείται και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι δεν λειτουργεί στα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μα αυτό πήρε πάρα πολύ καιρό. Και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να το αξιοποιούμε όχι μόνο για να δίνουμε κατευθύνσεις και συστάσεις στις χώρες για τα μακροοικονομικά τους, αλλά και για την εφαρμογή και υλοποίηση ε, των οδηγιών. Αυτό θα βοηθήσει στη διαφάνεια και χρειαζόμαστε τέτοιες ανακοινώσεις όπως αυτή για την οδηγία των υπηρεσιών νωρίτερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο ε, σημεία και να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πρώτον, Έφυγε τώρα δυστυχώ η κυρία Βερνιό για την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσώνων. Τα κράτη-μέλη επικαλούνται την επικουρικότητα. Προσοχή εκεί. Είναι πολλοί υπάλληλοι, ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία και στη Γερμανία που φοβούνται μήπως τους αφαιρέσουμε την ανεξαρτησία τους. Μα είναι εσωτερική αγορά, ενιαία, δεν μπορεί τα κράτη-μέλη, όπως είδαμε στην Ελλάδα, να ε, βεβαιούν τα ίδια ότι όλα βαίνουν καλώς και είμαστε εντάξει. Εκεί χρειάζεται επίσης σωστή επικοινωνία. Ε, μια ερώτηση που με πιέζει. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε τα κράτη να μπορέσουν να εφαρμόζουν σωστά αυτές τις πολιτικές για την εσωτερική αγορά Πού αποφασίζονται στο Συμβούλιο δημοκρατικά από όλου του υπουργού, πώ μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επικοινωνία, στην ενημέρωση για τη σωστή εφαρμογή επιτόπου, γιατί επήγε αυτό το πράγμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε. Ε, θα ήθελα, επειδή πιέζει και ο χρόνος τώρα, να πω κάτι συγκεκριμένο χωρίς να κάνω γενικές αναφορές. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας βοηθήσετε σε δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, η περιβόητη, για να μην πω διαβόητη συζήτηση για τις εκχωρήσεις ή τις αναθέσεις. Γράφει ε, στην εισαγωγή ότι πάνω από 25 είναι οι αποφάσεις του ΔΕΚ που δείχνουν ότι το πρωτογενές δίκαιο δεν αρκεί αλλά επίσης ε, καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα δεν γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται. Αν είναι σωστοί οι ορισμοί ίδιοι για αυτά τα concessions. Και στην πρόταση που μας έχετε καταθέσει ε, δεν είναι ε, λιμένο το θέμα των ορισμών και του πεδίου εφαρμογής. Δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα μέσα σε ένα λεπτό, αλλά να το κοιτάξετε παρακαλώ στις υπηρεσίε σα. Μήπω πρέπει να διευκρινιστεί αυτό για ποιου τομεί και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή. Παράκληση, δεν θέλω απάντηση. Και ένα δεύτερο, για την ανάθεση ε, στους διαγωνισμούς σε τρίτες χώρε. Η αμοιβαιότητα είναι μια ιστορία πάρα πολύ περίπλοκη. Έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μείονεκτήματα. Ξέρω ότι αυτή την αρχή την έχουμε χρησιμοποιήσει ως προειδοποίηση ε, στις ε, στρατιωτικές προμήθειες αμυντικού υλικού. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε μετά το καλοκαίρι, έτσι όχι σήμερα, μετά τις διακοπές, ποιες είναι οι εμπειρίες που έχετε ήδη κάνει με αυτή την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των εξοπλισμών και αυτά τρίτες χώρες είναι. Παρακαλώ μην μου απαντήσετε τώρα αν θέλετε το Σεπτέμβριο. Okay. Ναι, ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξή σας για να ετοιμαστεί πριν το Σεπτέμβριο. Θα δείτε όμως εάν θα κατευθεί αυτή η υπόσχεση τον την 1η Σεπτεμβρίου ε, για την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, ε, κύριε Πρόεδρε, αλλά όπω είναι τόσο ευφύ οι συνάδελφοι, όλα έχουν καλυφθεί. Απλώ ήθελα να απευθυνθώ στον Επίτροπο και να μιλήσω για την οδηγία των υπηρεσιών και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Για τα διπλώματα ιδίω, ξέρω ότι ε, και η αξιοπιστία σα είναι μεγάλη και το κύριο σα, ώστε να δώσετε στα κράτη να καταλάβουν ότι για μα είναι τελείω αδύνατο να εξηγήσουμε στι επιχειρήσει μόνο στην Ευρώπη ότι ένα εύκολο και απλό μέσο που δεν έχει και μεγάλο κόστο, μάλιστα ε, βιώσιμο, μακροπρόθεσμο για να περιοριστεί το κόστος της ανάπτυξης δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται γιατί υπάρχει ένας τσακωμός. Είναι στη δική σας τη σοφία να καταφέρετε να περάσει το μήνυμα και σε εσά υπολογίζουμε το ίδιο ε, και για το θέμα της εσωτερικής αγορά και των κοινωνικών δικαιωμάτων τη κοινωνική Ευρώπη. Καλώ ήρθε και ο κ. Ντεγιόνγκ ανάμεσα στου φίλου τη εσωτερική αγορά. Να μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα τη Ευρώπη είναι αντιαγωνιστικότητα. Ο καλύτερο τρόπο να αγωνιστούμε κατά τη ανεργία και να δώσουμε δουλειά στα παιδιά μα είναι ακριβώ να δώσουμε τη δυνατότητα στι επιχειρήσει μα να προσλαμβάνουν ανθρώπου. Διότι, κύριε Ντεγιόνγκ, κυρία Γκέπχαρτ, μπορούμε να περιλάβουμε στα κείμενά μα όσο θέλουμε την κοινωνική Ευρώπη, τα κοινωνικά δικαιώματα, ό,τι μα αρέσει. Εντάξει, προσυπογράφω κι εγώ. Όμω δεν θα υπάρξει δουλειά έτσι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στις επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι ότι σε εσά υπολογίζουμε για να ανακάμψει η απασχόληση και η ανάπτυξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς ό,τι μπορούμε για να αρθούν οι φραγμοί, τα σύνορα, τα εμπόδια. Και Γι' αυτό θα πρέπει το μήνυμα αυτό να είναι πολύ ηχηρό αυτή τη στιγμή. Όλοι κάνουν λόγο για ανάπτυξη. Ακόμη όμω στο κέντρο τη ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει τεθεί η εναρμόνιση ε, τη εσωτερική αγορά. Επιπλέον μιλάμε για μια τεράστια ε, κοινωνική οικονομική μάλλον δομή. Και αυτά ενώ κινδυνεύουμε να έχουμε δύο ευρωζώνες, τη μία που ασθενεί και την άλλη που υγιένει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σκεφτούμε για ποιους θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την αγορά. Για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, αλλά και επιχειρήσεις είναι ε, καταναλωτές. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, εδώ υπολογίζουμε σε εσά για να περάσει αυτό το καθοριστική σημασία πολιτικό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Και μιλήσατε και για χειροπιαστά θέματα. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ και η ενεργητικότητά σας και σας συγχαίρω, σα ευχαριστώ που δεν δείχνεται ε, ανοχή για την έλλειψη και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Πραγματικά, στη διακυβερνητική λύση πιστεύετε ότι μπορεί να ασκηθεί πίεση ώστε τα κράτη-μέλη να πιεστούν, να υλοποιηθούν όσα ήδη υφίστανται νομοθετικώς. Έπειτα, να σας ευχαριστήσω και λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ, που μιλήσατε για το πρόγραμμα δράσης για το εμπόριο και που το έχετε συμπεριλάβει στη δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσωπική σας στράτευση για το θέμα αυτό και τα όσα κάνουν οι υπηρεσίες σας για το πρόγραμμα δράση για το εμπόριο. Η 4η Ιουλίου είναι σημαντική ημερομηνία, το ξέρετε κι εσείς, αλλά ακριβώς τότε ο διάλογος για την πρωτοβουλία αυτή βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων θα οδηγήσει στην παρουσίαση εφαρμοστικών μέτρων. Είναι τεράστια η πρόκληση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι στις δυνάμεις μας, ώστε οι Βρυξέλλες να περάσουν σε όλη την αλυσίδα διανομής, να περάσουν μέχρι τους καταναλωτές οι κανόνες μας. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά ως τελευταία ρίψω κινδύνεψα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πολύ σύντομα γιατί πρέπει να συναντήσω τους εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στα πλαίσια της αμοιβαιότητας. Απλώς ε, συνεχίζοντας την παρέμβαση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ, ναι και εγώ προσέχω ιδιαίτερος και περιμένω να δω τι θα γίνει στις 4 Ιουλίου. Προτιμώ και εγώ την επίτευξη συμφωνίας και όχι τον ε, φραγμό και τη δυσκολία. Είναι η πρώτη μου αντίδραση αυτή, επειδή έχω κολλήσει. Το έχω πει άλλωστε και με την αφορμή τη οδηγία ε, για τι υπηρεσίε πήγα να συναντήσω όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών οργάνωσα ε, εργαστήρια με 800 ε, εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους. Κύριε Σφάμπ, ε, ρωτήσατε τι πρέπει να γίνει για να πετύχουμε να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και να μην οφαλοσκοπούμε ή να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς μπορούμε να κάνουμε μέσω των Υπουργών, μέσω των Εθνικών Βουλευτών. Πρέπει να συναντιόμαστε. Αλλά και οι Εθνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι. Πρέπει και εκείνου να του συναντούμε, να του σεβόμαστε, να του κάνουμε να συμμετέχουν. Έτσι έγινε με αυτή την ομάδα δράση των 800 υπαλλήλων που ασχολήθηκαν με όλα τα θέματα τη εσωτερική αγορά. Του συνάντησα προσωπικά και του ενημερώνα για τι συζητήσει μα. Όμω, ε, πολύ σωστά το είπατε αυτό, κυρία Κοράτσα Χρειάζεται η αυτορύθμιση. Σύμβαση λοιπόν, συμβόλαιο, συμφωνία προοπτική λύση των προβλημάτων από τους φορείς του ίδιου του κλάδου. Θα φροντίσω να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και ο μηχανισμός να λειτουργεί. Και εδώ θα μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνε. Και θα το κάνουμε ως δι. Ο κύριος Σβάμπ μίλησε για επικοινωνία ανέκαθεν πίστευα ότι πρέπει κανείς να ενεργεί αλλά και να ενημερώνει για αυτά που έχουν ήδη γίνει. Δεν μπορούμε να ενημερώνουμε για κάτι που δεν έγινε. Έχουμε ασχοληθεί με όλους τους τομείς, τώρα θα αρχίσουμε να συζητούμε, να συνεννούμαστε, όχι όπως έκανε πάντοτε η Επιτροπή top-down, από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά και αντιστρόφως. Ε, ελπίζω ιδιαιτέρως ότι η εβδομάδα για την ενία αγορά, όπως οργανώθηκε, θα μπορούσε να οργανωθεί με μια εβδομάδα ίσω για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλη μία, 15 ε, έως 22 Οκτωβρίου, για την εσωτερική αγορά και με συμμετοχή όλων των μέσων επικοινωνία που διαθέτουμε για να δούμε τι επιτυχίε, τα δυνατά σημεία, τι αδυναμίε τη εσωτερική αγορά. Να ξεφύγουμε από το πλαίσιο συνεδριάσεων που βρισκόμαστε μόνο μεταξύ μα και να δούμε ακριβώ τι έχουν να πούνε και οι πλογοί στο διαδίκτυο. Ήδη 200 άτομα έχουν εγγραφεί στον ιστοτοπό μα από τα 27 κράτη-μέλη. 200 μάλλον εκδηλώσει κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα για την εσωτερική αγορά θα συνεχίσουν να αυξάνονται, πιστεύω. Όπω είπα και στι δύο ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα δείξουμε πίκια για την ε, κακή υλοποίηση των κειμένων, για τι υπηρεσίε για την εσωτερική αγορά. Έχω ακούσει τις εξηγήσει, έχω καταλάβει τις δικαιολογίε, αλλά θα επιταχύνουμε το ρυθμό. Όπως είπε ο κύριος Σφάμπ, θα οδεύσουμε προς την μηδενική ανοχή. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν οι πίνακες αντιστοιχήσεις. Νομίζω ότι είναι απαραίτητοι το κείμενο των δικτών, benchmarking, για να δούμε ποιος κάνει τι στην Ευρώπη και θα δείτε και τα αποτελέσματα, διότι όσοι έχουν καλούς βαθμούς ή κακούς βαθμούς θα είναι πλέον γνωστοί. Και υπάρχει ένα εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα. Το αναφέρατε για την εσωτερική αγορά. Είναι πια το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει και αυτό να αξιοποιηθεί για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην εσωτερική αγορά. Σημείωσα τις παρατηρήσεις της κυρίας Βάιλερ Παρόλο που με συμβουλέψατε να μην σας απαντήσω, εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Και συμφωνώ μαζί σας, η νομολογία του ΔΕΚ, όπως την αναφέρατε, δεν προσφέρει από μόνο της αρκή νομική βεβαιότητα. Συμφωνώ επίσης, με όσο είπε ο κ. Ζιβά, ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογής της πρότασης για τις εκχωρήσεις. Ιδίω για ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την συνεργασία δημόσιο τομέα με δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς ε, θα μπορέσει να εφαρμοστεί το κείμενο αυτό. Και απειχώντας και προσπαθώ να συμφιλειώσω διαφορετικές απόψει αυτές τη κυρία Κοράτσα Μπίλτ με συναδέλφου τη άλλων ομάδων, Απηχώντας λοιπόν αυτές τις απόψεις, να πω ότι η ανταγωνιστικότητα έχει αξία και για τις περιοχές της Ευρώπης και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα άτομα. Δηλαδή, όταν είναι κανείς νέος και ξέρει πολλές γλώσσες και έχει μια διαβίου κατάρτιση, υπάρχει εδώ και το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, της προσωπικής ανταγωνιστικότητας. Επίσης, κυρία Κοράτσα Μπίλτ, νομίζω ότι χρειάζεται βιώσιμη οικονομική αποδοτικότητα της ε, ενιαίας αγοράς. και για την κοινοτομία και για την κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται κοινωνική συνοχή και μέσα στι επιχειρήσει αλλά και στον κοινωνικό ιστό γενικότερα. Κοινωνία χωρίς ε, κοινωνική συνοχή είναι κατακαιρματισμένη, είναι διχασμένη. Πέραν λοιπόν των κειμένων που είναι αυστηρά και πρέπει να τα σέβεται κανείς όπως με το άρθρο 1 της Οδηγίας Υπηρεσιών, υπάρχουν εργαλεία, αλλά μου κάνει εντύπωση η απήχηση που είχε η ευρωπαϊκή αυτή πρόταση από τους κοινωνικούς εταίρους και τους επιχειρηματίες. Σε όλη την Ευρώπη τώρα ξεκινούν να συζητιούνται ιδέες, ε, απόψεις που ξεκίνησαν με την Ευρωπαϊκή μας πλατφόρμα, αυτή της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γνωστό πια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά και μιλάμε για εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ανταγωνιστικό τομέα, για ε, επιχειρήσεις επικερδής που είτε έχουν διοντολογική οργάνωση αλληλέγγυα ή προσπαθούν να κατακτήσουν νέα μερίδια αγοράς. Ίσως και οι δύο αυτές πορείες να είναι παράλληλες. Είναι λοιπόν και αυτός ο τομέας σημαντικός. μας συγχωρείτε που μακρηγόρησα και σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την ε, προσοχή σας. Well, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που πάτε. Δεν σας είπα ότι λύεται η συνεδρίαση. Ξέρω ότι πεινάτε, αλλά σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι πεινάτε, αλλά έτσι δεν είναι πολύ κομψό και ευγενικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματός σας ε, τον Επίτροπο ε, που ήταν πραγματικά άθλος ε, αυτό που κατάφερε να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ήταν πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και διευρύναμε γενικά τη στρατηγική γύρω από ε, την ενία αγορά και από το 1992 έχουμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα, ε, μια στρατηγική να προωθήσουμε την ενιαία αγορά. Πολλά ε, έχουν γίνει χάρη σε εσά, αλλά και χάρη στη συνεργασία μας. Και ακριβώς αυτό είναι η αγορά, μια ενιαία ε, ολοκληρωμένη συνολική αγορά για τους πολίτες, καταναλωτές, εταιρείες, επιχειρήσεις. Και αυτό κυριάρχησε σήμερα στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ όπως πάντα που έρχεστε. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς ε, για τη μικρή υπέρβαση ωραρίου και θα το ξαναπούμε μετά τις διακοπές για τον επόμενο γύρο συζητήσεων για τη δεύτερη πλέον πράξη για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ.